Colleagues, good morning. Καλημέρα συνάδελφοι. Πριν πάμε στην ψηφοφορία, θα ήθελα να πω ότι έχουμε επισκέπτες από την Ρουμανία, από το Γκαλάτ, περιοχή της κυρία Τσικάου. Και έχουμε ευρωβουλευτή από το Ρουμανικό Κοινοβουλίο και κάποιους δημοσιογράφους. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Θα περιμένουμε την επόμενη ομάδα επισκεπτών. Έχουμε και άλλη ομάδα, θα έρθει αργότερα. Καλώ. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η ψηφοφορία όσον αφορά την έξι του κ. Μπράντμπον για το μέλλον των περιφερειακών αεροδρομίων και των υπηρεσιών. Έχετε πάρει όλοι τις κάρτες μαζί σας για την ψηφοφορία. Ναι. Ας κάνουμε έναν έλεγχο. Μια δοκιμή ψηφοφορίας, να δούμε πώς παραπάνω έχουμε το ΕΛΚ αυτή την εβδομάδα. Ξεκινά ε, η δοκιμή. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Και το ΕΛΚ είναι νόμιμο αυτή τη στιγμή. Είναι εντάξει. Okay. we'll start with... Ξεκινάμε με τη συμβιβαστική 4. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. we 12. είναι επόμενη υπέρ. Κάτα. Αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 8. Κατά τμήματα, ζήτησε το ECR. Πρώτο τμήμα. Έχει την άποψη. Λοιπόν, το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ή δεν ξέρω τι έκανε το ΕΛΚ. Ξεκινά λοιπόν ο έλεγχος. Η ψηφοφορία ηλεκτρονική. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά Αποχές εγκρίνεται. 43. Ρούμπικ. Σαν προστίκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 44. Το ίδιο προστίκι. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 48. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ρέτζι 3 κατά τμήματα πρώτο τμήμα καλή μέχρι πιο ελκυστικό Το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε. Το πρώτο καταπίπτει διότι εγκρίναμε την 47. Δεύτερο τμήμα. Σημειώνει ότι προγράμματα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 49. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 5 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος για τη Ρέτζι 5 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας και απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός ελέγχος της 51 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας Yeah. Can we close the vote now? Right. Vote is closed. And that's adopted. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Those against. Κατά. Έλεγχος για τα 52. Άρχεται η ψηφοφορία, ο έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. And that is adopted. Εγκρίνεται. 53 της υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές έλεγχος της 54 άρχεται η ψηφοφορία Everybody voted. Vote is closed. Πέρας Εγκρίνεται. Compromise 7. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 61 next Marinescu. 61 Μαρινέσκου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μπορείτε να σηκώνετε λίγο το χέρι πιο ψηλά, παρακαλώ. Κυρίως η ομάδα μου. Κάπως έτσι κουρασμένους τους βλέπω, δεν έχουν πολλή ενέργεια. Κοιτάω. Έτσι, σαν μαραμένο. 62. Σας όλοι. Υπέρ. Καλούς τους βλέπω τώρα. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 64. Λάιχφριντ. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε όλη την παράγραφο την, στην 68 υπέρ κατά αποχές έλεγχος της 68 άρχεται η ψηφοφορία. is closed. Πέρας. Rejected. Where do we go now? 66. Λοιπόν, μετά Λίχτεμπεργκερ κατά τμήματα, σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα το υπόλοιπο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 ένα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 μπαχ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ρέτζι 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 6 κατά τμήματα, το ζήτησε το ΕΛΚ, δύο τμήματα, μέχρι οικοδόμηση νέων, το πρώτο τμήμα, το... λοιπόν το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές έλεγχος του δεύτερου τμήματος, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 75 καταπίπτει. was accepted, so we still go to 76. Okay. 76. 76. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπό τον όρο ότι η Ιταλική εκδοχή είναι αυτή που γράφεται εδώ υπέρ ε, και διαβάζει Ιταλικά ο πρόεδρος θεωρώντας τα αεροδρόμια 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ελπίζουμε ότι ελπίζω να είναι σωστό το κείμενο, το ιταλικό 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 Λίχτεμπεργκερ υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη Ρέτζι 7 τώρα. Κατά τμήματα. Δύο τμήματα έχουμε. Μόνο το δεύτερο τμήμα. Το πρώτο τμήμα καταπίπτει διότι ψηφίσαμε συμβαστική 9. Ψηφίζουμε μόνο το δεύτερο τμήμα της Ρέτζι 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 93. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 106 τώρα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά σε ελέγξουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία 104 ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 107 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 καταπίπτει 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 καταπίπτει 105 Κατά πίπτη 114 υπέρ κατά αποχές ας γίνει ελέγχος για την 114 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ. 116 υπέρ κατά άποχες έλεγχος για την 116 νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά σε ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 117 Λίχτεμπεργκερ υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος 117 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι τέλος απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές ας γίνει ένας έλεγχος για την 122 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 123 έλεγχος. Ξεκινάει. Ψηφίσατε Τέλος. Εγκρίνεται. 125. Ρούμπιξ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά Όχι, δεν εγκρίθηκε 125. Λοιπόν, ξαναδοκιμάζουμε το 127. Ξανά από την αρχή, 127 υπέρ κατά αποχές έλεγχος νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά κάνουμε έναν έλεγχο ξεκινάει τώρα ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται 128-129 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Ρέτζι 10. Ρέτζι 10 αν παρακολουθείτε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 144 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 145 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος της 145, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας απορρίπτεται ε, στη ισοψηφία. 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 150 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 150 σας παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Κα... Απορρίπτεται με μικρή διαφορά. 151 σας όλοι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έχουμε τη συμβαστική, συμβιβαστική 1 με προφορική τροπολογία που ζήτησε το ΕΛΚ ποιος θα πάρει το λόγο ο κύριος Σασόλη είμαι αντίθετος με την προφορική τροπολογία Μπορείτε να το επαναλάβετε, λέει ο Πρόεδρος. Είμαι κατά αυτής τη προφορική τροπολογία. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδικασία. Έχετε αντίρρηση όσον αφορά την προφορική τροπολογία, λέει ο Πρόεδρος. Σε αυτή αυτή περιπτώση δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία, αλλά συμβαστική ένα χωρί την προφορική τροπολογία ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 Λίχτεμπεργκερ υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά κάνουμε έναν έλεγχο για τη 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 λέει ο πρόεδρος 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 27 άρχεται η ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται ε, με ισοψηφία. 30 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται 32 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 39 υπέρ, 3 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Μπράντμπερν. Next. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Next is Mr. Έκθεση του κυρίου Καντσιάν για τη χρηματοδότηση κοινωνικής συνδρομής προγράμματα καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας 2007-2013 και διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς και ενέργειας. Τροπολογίες 17 και 19 από κοινού. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 18. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 και 22. Με προφορική τροπολογία για την 22. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία. Όχι, οπότε τις ψηφίζουμε με την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 21. Ποιος είναι υπέρ.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 3 με προφορική τροπολογία. Έχετε αντιρρήσει. Όχι. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 ως προσθήκη υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για την τροπολογία 13 ως προσθήκη στην 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Everybody voted. Vote is closed. And that's rejected. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Everybody voted. Ψηφίσατε όλοι. Everybody voted. Last year. Τελευταία ευκαιρία παρακαλώ όσοι δεν ψήφισαν. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 35 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 3 αποχές. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια στον κύριο Κάντσιαν. Have we got the budget rapporteur here yet? Just checking on whether the general budget rapporteur has arrived. Περιμένουμε τον εισηγητή μας για τον προϋπολογισμό του 2013, τον γενικό εισηγητή.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 Ευχαριστώ. Okay, colleagues. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ας επαναλάβουμε τη συνεδρίαση. Καλώς ήρθατε κύριε Γενικά, Γενική, Γενική για τον προϋπολογισμό. Κύριε Λαβία, η Επιτροπή μας είναι από τις καλύτερες Επιτροπές του Κοινοβουλίου και κυρίως αν μας δώσετε κάμποσα δισεκατομμύρια ευρώ ε, θα είμαστε οι καλύτεροι φίλοι σας. Αλλά ίσως εσείς θα μας εξηγήσετε τώρα το σενάριο για τον γενικό προϋπολογισμό. Έτσι ε, σας δίνω το λόγο αμέσω και καλώς ήρθατε και πάλι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συμμετάσχω σε αυτή την συνάντηση με την Επιτροπή Μεταφορών. Ε, Ήρθα σε επαφή με τον Γενικό Εισηγητή Υπολογισμού να πω ποια διαδρομή θα ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στον ορισμό του προπολογισμού. Απ' την άλλη πλευρά, ποιε είναι οι κατευθυντήριε γραμμέ που έχουμε εγκρίνει ε, Λοιπόν, επαναλαμβάνω συντομία. Μέσω αυτών των συναντήσεων με τις ειδικέ επιτροπές, αρμόδιες επιτροπές, θέλουμε να έχουμε άμεση επαφή που μπορεί να μας επιτρέψει, να επιτρέψει σε όλους να αισθανθούν ότι είναι τμήμα της διαδικασίας της λήψης ε, απόφασης για την κατάρτιση του προπολογισμού του 2013. Όπως θα σημειώσω το 2013 είναι το τελευταίο έτος των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013. Και όπως συμβαίνει συχνά όταν υπάρχουν πολυετή προγράμματα, όπως είναι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην αρχή της περίοδου προγραμματισμού αναλαμβάνονται οι υποχρεώσεις και μετά όσο προχωράμε έχουμε τις ε, πληρωμές που καταβάλλονται. Είναι σαφές λοιπόν ότι σήμερα βρισκόμαστε το τελευταίο έτος του πολιτού πλαισίου για το 2013 και τον προπολογισμό αυτό έχουμε μεγάλη ανάγκη καταβολής πληρωμών το γνωρίζει όποιος συμμετέχει στην Επιτροπή Προπολογισμών ότι οι αιτήσει για πληρωμές με κάθε χρόνο αυξάνονται όσον αφορά την αύξηση της εκτελέσεις των προγραμμάτων, διότι πολλά κοινοτικά προγράμματα έχουν δρομολογηθεί και έχουμε μεγάλη ανάγκη πληρωμών. Αλλά αυτό έρχεται σε αντίθεση με την οικονομική αυτή τη μεγάλη κρίση. Ε, έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι πολλά κράτη-μέλη που δεν έχουν πλήρη αντίληψη του πώς λειτουργεί ένα πολιτές πρόγραμμα και πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και την ανάγκη πληρωμών που έχουμε, στο τέλος λοιπόν τα κράτη-μέλη έχουν την τάση να μειώνουν τις πληρωμές και τη δυνατότητα να έχει ένα επίπεδο πληρωμών επαρκέ ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Γι' αυτό στο τέλο του περσινού έτου έχουμε αιτήσει από τα κράτη-μέλη για πληρωμέ για 15 δισεκατομμύρια ευρώ ε, μόνο εν μέρη εκτελεστήσεις διότι δεν υπήρχαν επαρκείς δόσεις που κατεβλήθησαν πληρωμές. Όποιος ξέρει, όποιος είναι παρόν στην Επιτροπή Προπολογισμών, την περασμένη εβδομάδα ακούσαμε ε, μία έκθεση όσον αφορά τις περιφερειακές πολιτικές και εκεί διεφαίνεται, υπογραμμιζόταν ότι πολλά προγράμματα πολλών κρατών μελών δεν εδώ και πολλούς μήνες δεν δέχονται πληρωμές. Δεν ε, λαμβάνουν πληρωμές, γιατί δεν υπάρχουν επαρκή σπόροι. Λοιπόν, έκανα το γύρο των διαφόρων αρμοδίων ε, ε, επιτροπών. Κάνω αυτό το γύρο εν ώψη του 2013, διότι θα ήθελα να γνωρίζουν οι διάφορες επιτροπές, οι συνάδελφοι, ποια είναι η κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ώστε να μπορέσουμε να καταρτήσουμε ε, τον επόμενο προϋπολογισμό για το τελευταίο έτος των δημοσιονομικών προοπτικών. Ε, ετοιμάσαμε κατευθυντήριες γραμμές που είναι αρκετές, αρκετά γενικές. Ε, δεν μπήκαμε στις διάφορες προτεραιότητες των διαφόρων επιτροπών και θέλουμε να συμμετάσχουν όλες οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στον καθορισμό των προτεραιοτήτων των διαφόρων κονδυλίων εντός ενός πλαισίου με προτεραιότητες που έχει δημιουργηθεί. Η γενική προτεραιότητα είναι από την πλευρά η ανάπτυξη και από την άλλη η απασχόληση με ιδιαίτερη αναφορά στην απασχόληση των νέων. Αλλά η ανάπτυξη και ε, η απασχόληση εξαρτώνται από διάφορε γραμμέ του προπολογισμού και γι' αυτό χρειάζεται η συνεργασία των διαφόρων επιτροπών που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και πολύ καλύτερα προφανώς από το Γενικό Εισηγητή ε, σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα προγράμματα, ποιες είναι οι ανάγκες και ποιες δυνατότητες ε, υπάρχουν αυτές οι γραμμές να μπορέσουν να συμβάλλουν στη γενική στρατηγική που θέλει να εφαρμοστεί. Είναι σαφές ότι κάθε επιτροπή και συνήθως το Κοινοβούλιο ζητά κάτι περισσότερο, κάτι περισσότερο για τα κονδύλια τα οποία υπάρχουν και εκεί που κινείται η Επιτροπή, συγκεκριμένες γραμμές του προπολογισμού για κάθε Επιτροπή. Χρειαζόμαστε όμω ένα πλαίσιο λιτότητα γενικό που επικρατεί και σε γενικέ οικονομικέ δυσκολίε να ζητήσουμε από τι επιτροπέ όχι μόνο να εντοπίσουν τι προτεραιότητε τι θετικέ, τι προτεραιότητε επί των οποίων θα πρέπει να επικεντρωθούν οι πόροι, αλλά να μα πούν κατά πόσο υπάρχουν κάποιε γραμμέ του προπολογισμού ε, που δεν έχουν επίπεδα σε επαρκή, κονδύλια ή προγράμματα που δεν δαπανούν σύμφωνα με τι προβλέψει ε, τα χρήματα, ούτως ώστε ίσως να, να ε, προγραμματίσουμε αυτές τις γραμμές. Άρα χρειάζομαστε οι διάφορες επιτροπές στα πλαίσια και του τριμερούς διαλόγου και στις διάφορε διαδικασίε του προπολογισμού να εντοπίσουν όχι μόνο τι θετικέ προτεραιότητες, αλλά και τι αρνητικέ, και αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα ευθύνη που θέλουμε να στείλουμε ε, ως κοινοβούλιο. Ένα άλλο θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι καλό να το υπογραμμίσω και σα το αναφέρω είναι των διαφόρων πιλωτικών προγραμμάτων, των προπαρασκευαστικών δράσεων, ε, διότι είναι από τις προτεραιότητες που παραδοσιακά ε, έχει το Κοινοβούλιο και περνάμε και μια συγκεκριμένη διαδρομή. Λοιπόν, ζητούμε τα διάφορα πιλωτικά προγράμματα και παρασκευαστικέ δράσεις να παρουσιάζονται στις επιτροπές και από τις επιτροπέ στην Επιτροπή Προπολογισμού μετά μέχρι το τέλος του Μαΐου, ούτω ώστε τις αρχές του Ιουνίου να μπορέσουμε να αποστείλουμε αυτή την πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνει μια αρχική εκτίμηση της δυνατότητα εκτελέσεως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά να βάλουμε στο πακέτο το τελικό που θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών και θα ψηφίσουμε στο Κοινοβούλιο μόνο ε, αυτά που μπορούν να εφαρμοστούν τόσο να χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους λίγους πόρους που διαθέτουμε. Ε, είναι σαφές ότι από εδώ μέχρι τη στιγμή που θα εγκρίνουμε τον προπολογισμό ε, έχουμε μια διαδρομή που θα πρέπει να διατρέξουμε και θα ξεκινήσουμε την εξέταση της ε, πρότασης που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει στις 25 Απριλίου όπου εκεί θα τονίσει και υπογραμμίσει τι ανάγκε από πλευρά αναλήψεω υποχρεώσεων και πληρωμών για κάθε γραμμή του προπολογισμού. Ξεκινώντα από εκεί, θα, θα κάνουμε τι δικέ μα σκέψει και εξετάσει, επειδή διάφορε επιτροπέ θα τοποθετηθούν και θα αναπτύξουμε μία πορεία που θα μα οδηγήσει, ελπίζω, στο τέλο του έτου, μετά από τη συνδιαλλαγή, να έχουμε έναν προϋπολογισμό εγκεκριμένο στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Thank Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λαβία. Ο κύριος Ρίκε. Α, ναι, συγγνώμη. Εσείς η κυρία Μάισνερ. Δεν πειράζει. Ο Ντομινίκ είναι γνωστόν άλλωστε ότι ασχολείται με τον προϋπολογισμό. Εγώ λιγότερο γνωστή. Ευχαριστώ λοιπόν πρώτα τον κύριο Λαβία που ήλθε να μα απευθύνει τον λόγο. Πρόκειται για νέα διαδικασία και εγώ τη βρίσκω καλή σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό. Το κοινοβούλιο είναι αρκετά ενωμένο. Βέβαια η Επιτροπή προπολογισμών, κάπω υπερίπταται όλων των υπολείπων και λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ολόκληρου του Κοινοβουλίου, ενώ οι επιμέρου επιτροπέ προσπαθούν να προωθήσουν τα δικά του θέματα. Αυτό είναι σαφέ για μένα. Γενικά, ωστόσο, θεωρώ και καλά τα εξηγήσατε. Είναι κατανοητό ότι οι χώρες μέλη θέλουν να προχωρήσουν σε περικοπές, διότι θέλουμε βέβαια Ευρωπαϊκή Ένωση σταθερότητας, βελτίωση των δημοσιονομικών συνθήκων και στις χώρες μέλη και εάν από την άλλη μεριά αυξάνουμε τις δαπάνες θα είναι παράλογο. Δηλαδή δεν θα μπορούν να πληρώσουν πλέον οι χώρες μέλη. Έτσι λοιπόν δικό μας καθήκον είναι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπερασπιστούμε τον ενωσιακό προϋπολογισμό, διότι όπως είναι, είναι μας είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Διότι και παραπάνω χώρες μέλη έχουμε πλέον, άλλωστε θα προσθεθεί άλλη μία, αλλά και έχουμε και περισσότερες αρμοδιότητες. Δηλαδή και οι προσδοκίες... απέναντί μα μας είναι μεγαλύτερες. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε περίκοπες... λοιπόν υπό την έννοια αυτή. Ελπίζω ότι όλοι θα μείνουμε ενωμένοι. Ότι εν μέρη δεν απορροφώνται όλα τα κονδύλια το γνωρίζουμε. Μιλήσατε για τις σχετικές πολιτικές. Σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, για παράδειγμα, ήδη μιλήσαμε στις πιο πρόσφατες ημέρες αφιερωμένες στα ε, διευρωπαϊκά δίκτυα. Είπαμε με το αγγλικό εκείνο «use it or lose it» και για τις μεταφορές στην Ευρώπη δεν έχει νόημα να, είμαστε, να γεμίσουμε την Ευρώπη εργοτάξια που δεν τελειώνουν ποτέ δεν προσφέρει αυτό καμία ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Άρα και εδώ πρέπει να... Ε, εδώ και εδώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Σήμερα είχαμε μια πρώτη συνάντηση με ένα σκιώδη συγητή, τον οποίο προσεκάλεσα εγώ, και αυτό υπογραμμίσαμε ιδίω ότι είναι σωστό να γνωρίζουμε, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, που εντοπίζονται κονδύλια τα οποία δεν έχουν αναρωθεί. Αυτό θα εξυπηρετήσει άλλωστε και τη στρατηγική Ευρώπη 2020, διότι ανάπτυξη και απασχόληση είναι κάτι το οποίο απασχολεί και εμάς, τις ειδικέ επιτροπές. Και για τα πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικά μέτρα, προς αυτή την κατεύθυνση θα κάνουμε προτάσεις. Εξηγήσατε και το χρονοδιάγραμμα, το οποίο και εμεί το συζητήσαμε σήμερα το πρωί. Θα περιμένουμε πρώτα λοιπόν τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ μπορώ να πω λίγα πράγματα. Δηλαδή, πέρσι από τι χώρε μέλη έγιναν περικοπές στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς των μεταφορών και με κοινή ψήφο στην ε, Επιτροπή Προϋπολογισμών καταφέραμε να ανατρέψουμε τις περικοπές αυτές, διότι εν τέλει οι οργανισμοί αυτοί έχουν αναλάβει περισσότερα καθήκοντα. Δεν μπορούμε να τους περικόπτουμε τα κονδύλια. Κάτι άλλο το οποίο θέλω να τονίσω και πάλι είναι ότι έχουμε αρμοδιότητα και για τον τουρισμό με την ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Και μέχρι τώρα για τον τουρισμό έχουμε μόνο προπαρασκευαστικά μέτρα, τα οποία έχουμε βέβαια εγγράψει στον προπολογισμό, δεν, έχει όμως, δεν υπάρχει όμως ακόμα σχετικός τίτλος. Και επιθυμούμε και ε, προσπαθούμε να επιτύχουμε να περιληφθεί και ειδικό τίτλος. Διότι δεν έχει αλλιώς νόημα να έχουμε αρμοδιότητα και να είμαστε υποχρεωμένοι να βγαίνουμε στη ζητιανιά για τα απαραίτητα κονδύλια για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες της αρμοδιότητας αυτής. Υπάρχουν βέβαια και πολλά άλλα έργα. Ένα μόνο τελευταίο σχόλιο θα κάνω όμως. Η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Αυτή δεν αφορά μόνο τη δική μας Επιτροπή αλλά και άλλες. Και γνωρίζουμε ότι για αυτή τη διευκόλυνση προτάθηκαν 50, 50 δις και γνωρίζουμε επίση ότι οι χώρες μέλη θέλουν να κάνουν περικοπές σημαντικές στον τομέα αυτό. Εγώ το προσέχω ιδιαίτερα αυτό και θα συνεχίσω να το προσέχω, αλλά καθώς και άλλα μέλη τη Επιτροπής μα, διότι αφενός υπάρχει η φάση των πιλωτικών προγραμμάτων η οποία ε, λειτουργεί ήδη από φέτος και όπου προσπαθούμε να επιτύχουμε την προσέλκυση και ιδιωτικών κεφαλαίων, προσφέροντας δηλαδή και κεφάλαια της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και για του χρόνου θα χρειαστούμε κάποια κονδύλια για να προπαρασκευαστεί η φάση του συνδέοντα στην Ευρώπη. Και αυτά λοιπόν θα τα υποβάλουμε ως προτάσεις εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, τη δική σας δηλαδή. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι που ήλθατε και θα συνεχίσω με τη συνεργασία μαζί σας όπως έχει αυτή άλλωστε ε, ισχύσει και τα τελευταία χρόνια με την ελπίδα ότι θα καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Για το Λαϊκό Κόμμα τώρα, ο κύριος Ρικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον ε, Γενικό Εισηγητή. Βρίσκω ότι είναι πολύ σημαντικό που ήρθατε γιατί μας δίνετε μια εικόνα γενική Βέβαια οι ειδικέ θεματικές επιτροπές πρόθουν τα δικά του ενδιαφέροντα. Θέλω να θέσω ορισμένα θέματα. Το πρώτο υπογραμμίστηκε και από τον Τζάνι. Υπάρχει ένα κενό 15 δισεκατομμυρίων στις πληρωμές που δεν κατόρθωσε ο προϋπολογισμός του 2011 να καλύψει το κόστος ορισμένων δράσεων στην περιφερειακή πολιτική. Το πρώτο που πρέπει να λεχθεί λοιπόν είναι ότι αυτό το κενό στις πληρωμές οφείλεται στο ότι δεν λειτουργήσε καλά η πολιτική, η περιφερειακή πολιτική, στο πλαίσιο το, και όταν θα αρχίσει μάλλον να οριμάζει το δημοσιονομικό πλαίσιο θα βελτιωθεί η κατάσταση. Για την πολιτική των μεταφορών τώρα, η οποία καταναλώνει τακτικά κονδύλια, υπάρχουν, υπάρχει το πρόβλημα ότι η κατανάλωση αυτή καλύπτει όλες τις ειδικέ επιτροπές. Τα 10 ή 15 δισεκατομμύρια των πληρωμών, των καθυστερούμενων πληρωμών από πέρσι, που θα επιβαρύνουν βέβαια τον προπολογισμό του 2012, αντιστοιχούν και σε πληρωμές οι οποίες δεν έγιναν και τα προηγούμενα χρόνια και επομένως επιστράφηκαν τα κονδύλια στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Άρα κάποια στιγμή έχασε τις πιστώσεις αυτές ο κοινοτικός προϋπολογισμός και πήγανε στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Τώρα βέβαια οι χώρες μέλη δεν έχουν την θέληση να ξαναβγάλουν τα χρήματα αυτά για το 2012. Τέλος, για τις πληρωμές το πρόβλημα των περιθωρίων για τον προϋπολογισμό του 2012 που θα είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Και αυτό θα βαρύνει ιδιαίτερα στα πιλωτικά προγράμματα και στις προπαρασκευαστικές δράσεις. Και είναι ακόμα πιο δύσκολο τότε το έργο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, διότι ο τουρισμός που αποτελεί τη νέα αρμοδιότητα της Ένωσης μέχρι τώρα δεν είχε στη διάθεσή του παρά μόνο τι πληρωμέ, δηλαδή για πληρωμέ των προπαρασκευαστικών δράσεων και πιλωτικών προγραμμάτων. Όπου ο προπολογισμό εκεί δεν είχε κάνει διάκριση σαφή για τον τουρισμό. Για, τις αυτές, για νέα αυτή αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου. Κάπου αυτό συμπιέστηκε στους δύο προηγούμενους προπολογισμού. Δεν περιλήφθη περιλήφθη δηλαδή ειδικά στον προπολισμό. Ούτε τώρα για το 2012 η εικόνα είναι πολύ καλή, διότι τα περιθώρια είναι πάρα πολύ περιορισμένα και αυτό θα έχει επιπτώσεις στις ε, προπαρασκευαστικές δράσεις και στα πιλωτικά προγράμματα. Αυτά για τις νέες αρμοδιότητες. Ελπίζω ότι δεν θα συμβεί το ίδιο με άλλες πολιτικές και το πρόβλημα των ε, οργανισμών είναι πολύ περίπλοκο για τις μεταφορές ιδιαίτερα δηλαδή. που βρίσκονται διαρκώς στο στόχαστο του Συμβουλίου οι οργανισμοί αυτοί με μείωση του προϋπολογισμού τους. Δύο πράγματα τα οποία είναι σημαντικά δηλαδή για μας. Οι νέες πολιτικές για τον τουρισμό και οι, εκτελεστικοί, και οι οργανισμοί όπως οι οργανισμοί που έλεγα πριν, αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν από περικοπέ. Το επισημαίνω αυτό στον εισηγητή, διότι μπορεί να έχει πολύ αρνητικέ συνέπειες για μας. Εν τέλει, δεν γνωρίζω ποια είναι η απορροφητικότητα των κονδυλίων στο επίπεδο του, των μεταφορών. Οι μεταφορές καταναλώνουν πολλά κονδύλια Και κύριε Σεγητά, συμφωνούμε με τις γενικές αυτές ανησυχίες του Κοινοβουλίου και ειδικότερα της Επιτροπής Προπολογισμών για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Οι μεταφορές είναι ένα αντικείμενο το οποίο που εντάσσεται στις ε, προηγούμενες, και στις προηγούμενες στρατηγικές ανέρχεται στο 10% του ΑΕΠ της Ένωσης και ένας παράγοντας πολύ σημαντικός για την ανταγωνιστικότητα. Που οφείλει να ενισχύσει και το, και το τωρινό δημοσιονομικό πλαίσιο. Δίνοντας επαρκή όθηση στην Επιτροπή Μεταφορών για να μπορέσει να πράξει τα δέοντα για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη. Thank you very much. Mrs. Ευχαριστώ. Από τους ε, δημοκρατικού, ε, δημοκρα... σοσιαλιστές δημοκρατικούς, κύριε Ρουμπιέρ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή αυτή η ιδέα ανάμειξη στη συζήτηση και στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όλων των ειδικών επιτροπών. Γιατί πολλές φορές ε, αυτές οι ειδικέ επιτροπές, οι δικευμένες επιτροπές ε, που επικεντρώνονται πολλές φορές στις πολιτικές που είναι αρμοδιότητάς τους, αλλά ξεχνούν μερικές φορές ότι όλες οι πολιτικές χρήζουν δημοσιονομικές υποστήριξης και αυτό δίνουμε να το ξεχνούμε εστιαζόμαστε μόνο στις δικές μας πολιτικές. Θυμόμαστε ότι για όλες μας τις προτεραιότητες χρειάζονται κονδύλια όταν φτάνει η ώρα της συζήτησης του προϋπολογισμού. Καλό είναι λοιπόν να μειγνύονται από νωρίς αυτή τη συζήτηση όλες οι ειδικευμένες επιτροπές. Και όσοι συμμετέχουμε και στην Επιτροπή Προπολογισμών, γνωρίζουμε ότι ο προπολογισμό και η διαπραγματεύση για τον προπολογισμό του 2013 θα είναι εξαιρετικά αντίξωε γιατί το 2013, όπως αναφέρθηκε, είναι η τελευταία χρονιά των αφισταμένων δημοσιονομικών προοπτικών. Τα περισσότερα ε, προγράμματα βαίνουν προς το τέλος τους, αλλά χρειάζονται συμπληρωματική χρηματοδότηση και λόγω των προβλημάτων ε, ε, χρηματοδότησης του 2011 και 2012. Οπότε έχουμε 11 δις πληρωμών από το 2011 που δεν έγιναν και μεταφέρθηκαν στο 2012 και τις προάλλες η Επιτροπή άρχισε ήδη να μας δίνει κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι και για το 2012 δεν θα έχουμε αρκετά κονδύλια. Οπότε θα πρέπει να προσφύγουμε σε διορθωτικούς προϋπολογισμούς. Επιπλέον μπαίνουμε σε προκαταρκτική φάση των διαπραγματεύσεων για, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και για τις ανάγκες της επόμενης επταετίας. Και φαίνεται ότι για μία ακόμη φορά το Συμβούλιο θα προσπίσει με νύχια και με δόντια περικοπές. Και φαίνεται ότι οι περικοπές θα έρθουν γύρω στα 200 δισεκατομμύρια. Πολύ περισσότερο δηλαδή από τον ετήσιο προϋπολογισμό μια, μιας χώρας. Γι' αυτό και θα χρειαστούμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών την αμέριστη υποστήριξη όλων των άλλων ε, ειδικευμένων επιτροπών. Θα πρέπει να συσπηρωθούμε και με μία φωνή να προσπίσουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί έρχονται πολύ δύσκολοι καιροί διαπραγματεύσεων, χαλεπές διαπραγματεύσεις, αν και θα είναι και ενδιαφέρουσες. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα της Επιτροπής σας, συζητήσαμε τις κατευθυντήρες γραμμές και το πρωί είχαμε μία πρώτη συνάντηση. Και όπως και στο παρελθόν η θέση της Επιτροπής Μεταφορών θα είναι ομόφωνη, αν και στις προκατακτικές δράσεις και στα πειραματικά σχέδια Υπάρχουν κάποια ζητήματα που με απασχολούν ιδιαίτερως. Καταρχήν το ελάχιστο περιθώριο που θα έχουμε στην σχετική κατηγορία ε, να βρούμε κονδύλια για να χρηματοδοτήσουμε τις δράσεις αυτές. Και το χειρότερο είναι ότι φαίνεται ότι χάνουμε το στόχο των προκαταρκτικών δράσεων και των πειραματικών ε, σχεδίων. Γιατί οι προκαταρκτικές δράσεις και τα πειραματικά σχέδια γίνονται για να δούμε αν οι ιδέες που ε, αναπτύσσουν είναι λειτουργικές και αν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε νέες πολιτικές. Αλλά φαίνεται ότι μετά από δύο-τρία χρόνια εφαρμογής το ξεχνάμε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να αναδείξουμε πυγμή απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πούμε ότι δεν επιτρέπεται αυτή η κατάσταση. Δεν μπορούμε κάθε δύο-τρία χρόνια να υποβάλλουμε νέες ιδέες και να ξεχνάμε τις παλιές. Δεν είναι αυτός ο στόχος ούτε των προκαταρκτικών δράσεων, ούτε των πειραματικών πιλωτικών σχεδίων. Για τον ε, βιώσιμο τουρισμό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει σε αυτό να επιμείνουμε. Περιμένουμε πάντως την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, που θα υποβληθεί την 25η Απριλίου. Πάντως φαντάζομαι ότι η θέση της ε, Επιτροπής Μεταφορών και στην περίπτωση αυτή θα είναι παρόμοια με τις προηγούμενες χρονιές. Πριν καλωσορίσω την κυρία Ντουιρόν των Πρασίνων, θα ήθελα να καλωσορίσω ε, μια ομάδα επισκεπτών από το Αβούργο Είναι προσκεκλημένη της κυρίας Μάισνερ. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω να απολαύσετε τη σύντομη διαμονή εδώ. Είμαστε σε ένα ε, ασήμαντο θέμα, όπως διαπιστώσατε, το θέμα της χρηματοδότησης. Καλημέρα σας πάντως και καλώς ήρθατε επισκέπτες από το Αβούργο. Η κυρία Ντιουρό από τους Πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες, γιατί έχουμε εδώ μέλη της Επιτροπής Μεταφορών και Επιτροπής Προϋπολογισμών. Για μένα το πρόβλημα είναι η τρύπα των 15 δισεκατομμυρίων, το πρόβλημα με τις πιστώσεις πληρωμών και γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα αυτά είναι ε, πολύ σημαντικά και πάντα Μα κρατάει ο μύρος στο Συμβούλιο με το πρόβλημα των πιστώσεων πληρωμών και με τις καθυστερήσεις που έχουμε θα αντιμετωπίσουμε και φέτος μεγάλες δυσκολίες. Στις, στην πρία των συζητήσεων για τη διαμόρφωση του προπολογισμού και στις διαπραγματεύσεις, στον τριμερή διάλογο δηλαδή με το Συμβούλιο, ε, θα πρέπει τα ομόλογα έργου να μην χρησιμοποιηθούν ως το νέο παιχνιδάκι, το καινούριο κοσκινάκι που θα μας καθυστερήσουν σε άλλες συζητήσεις. Συμφωνούμε και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ότι έχουμε περιορισμένα σχέδια, περιορισμένα ομόλογα έργου και όλοι συμφωνούμε γι' αυτό, αλλά δεν θα πρέπει να δώσουμε την ψευδέστηση ότι και άλλη χρηματοδότηση είναι δυνατή και ότι έτσι θα καθυστερήσουμε ακόμη περισσότερο σε ορισμένες πληρωμές. Κάτι άλλο που επίσης αναφέρθηκε, προσοχή ο προϋπολογισμός των μεταφορών να μην χρησιμοποιηθεί ως μεταβλητή προσαρμογής. Όταν ε, έχουμε περιθώριο χρηματοδοτούμε, όταν είναι ε, τσίμα τσίμα οι προϋπολογισμοί, από ποια κατηγορία αφαιρούμε, από τις μεταφορές. Όχι. Επίσης θέλουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία από τον εισηγητή για τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί βρισκόμαστε στο τελευταίο έτος του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Καλό θα ήταν λοιπόν να έχουμε ένα, μια επισκόπηση και των προηγούμενων ετών, ώστε να μπορούμε να προγραμματίσουμε το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διασύνδεση ε, με τον προπολογισμό του 2012, αλλά και με το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα πρέπει να συντονιστούμε με τον εισηγητή και με τα μέλη που συμμετέχουν και στις δύο επιτροπές για να εξασφαλίσουμε μια ευθυγράμμιση και παραλυσμό των σχέσεών μας, ώστε πραγματικά να προσπίσουμε ένα προπολογισμό ε, για τις μεταφορές αντάξιο του έργου μας. Ο κύριος Ζήλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να περιοριστώ σε λίγα θέματα, αυτά που εξετάζουμε για τις μεταφορές στα πλαίσια του προϋπολογισμού του 2013. Και να μην μιλήσουμε για τη γνωστή κατάσταση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη. Ποια θα είναι η κατάσταση του προπολογισμού του 2013. Σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, οι παρασκευαστικές δράσεις και τα πιλωτικά προγράμματα, γνωρίζουμε, όσοι έχουμε κάποια πείρα στα θέματα αυτά, ότι είναι κάπως τα παρατημένα παιδιά του προϋπολογισμού. Δεν θέλω να κοκολογήσω εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως, αν επικεντρωθούμε σε δύο-τρία πιλωτικά προγράμματα ή για προπαρασκευαστικές δράσεις για το 2013, θα πρέπει να δούμε πώς θα τα εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε καταρχήν ένα πρόγραμμα για τον τουρισμό, ένα για τις μεταφορές για να δούμε αν θα συνεχίσουμε αυτά τα πιλωτικά προγράμματα. Θα τα συνοδεύσουμε με νέα. Οι μεταρρυθμιστές συντηρητικοί δεν θέλουν αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για, τις, για τους οργανισμούς. Γιατί δεν είναι δυνατόν από τη μια να περιορίζουμε τους μισθούς μόνο στους εθνικούς προϋπολογισμούς και να ε, τους αφήνουμε άθικτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει στον προπολογισμό του 2013 να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, για, το, για, το, για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, για το Μάρκο Πόλο, το σύστημα ΣΕΖΑΡ και το ΣΕΖΑΡ για τις ε, επιχειρήσεις. Κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό για την ομάδα μου, τους μεταρρυθμιστές και συντηρητικού, είναι να διασφαλίσουμε τον προϋπολογισμό των μεταφορών και το 2013. Κύριος Φιντάντσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα να πω κάτι, διότι συμφωνώ απόλυτα και με τον συνάδελφο Μάισνερ και με τον Σκιώδη Ντομινίκ Να πω κάτι για την πολιτική του, του τουρισμού που αναφέρθηκε. Όταν ε, είναι σωστό αυτό που έλεγε ο Ντομινίκ σαν Επιτροπή Μεταφορών δεν ζητήσαμε γνωμοδότηση επί του προγράμματος Κόσμου όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ανήκει βασικά στην Επιτροπή Ήτρε, αλλά οι πόροι για τον τουρισμό στον προγραμματισμό 2014-2020 έχουν ενταχθεί εκεί. Είναι εντός μιας παραγράφου ειδική του κόσμου που προβλέπει ήδη σήμερα στην παρούσα πρόταση 131 εκατομμύρια ευρώ για ειδικά προγράμματα για τον τουρισμό. Και θέλω να κάνω το εξή αίτημα που ελπίζω να το υποστηρίζουν οι συνάδελφοι, τουλάχιστον εκείνοι που τοποθετήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ε, να επεξεργαστούμε εντός της Επιτροπής των Προϋπολογισμών ε, το θέμα και με την Επιτροπή ΣΥΤΡΕ να μπορέσουμε να εγκρίνουμε, να επιβεβαιώσουμε ότι θα δοθούν τα 131 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πρέπει να το θεωρήσουμε αυτό σαν έναν αριθμό που πρέπει να υποδιαιρεθεί σε 27 χώρες. Διότι θα είναι ψίχουλα έτσι, θα... αλλά θα είναι χρήσιμο αυτά τα χρήματα να αναπτύξουμε προγράμματα που δίνουν προστιθέμενη αξία ευρωπαϊκή και μπορούν να δώσουν συγκεκριμένη όθηση στον ανταγωνιστικότητα τουρισμού. Να εστιαστούμε ιδιαίτερα στο κομμάτι του κόσμου που αφορά την υποστήριξη των μικρομεσαίων ε, τουριστικών επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρινέσκου έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω στις και στους συναδέλφους της Επιτροπής Προπολογισμών ότι δεν πρόκειται μόνο για τον προπολογισμό του 2013 αλλά και του 2014 οι αριθμοί που θα, τα ποσά που θα καθοριστούν τώρα για το 2013 είναι πιθανόν εάν δεν συμφωνήσουμε για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να ισχύσουν και για το 2014. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο το καθήκον που έχετε αναλάβει. Και επιθυμώ να επισημάνω ότι στις διαπραγματεύσεις του περσινού χρόνου, τον Νοέμβριο του 2011, φάνηκε καθαρά ότι θα φτάσουμε στην κατάσταση το 2012 που περιγράφηκε πριν, ότι δεν είχαμε πλέον κονδύλια για τις πληρωμές. Και λόγω εσφαλμένων υπολογισμών από πλευρά κομισιών, θα θυμάστε ότι έλειπαν 1,5 δις ευρώ και λόγω της άρνησης του Συμβουλίου να διαθέσει πάνω από 500 εκατομμύρια. Έγινε έκθεση για διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2011 και στην κατάσταση αυτή φτάσαμε τελικά. Γι' αυτό και πρέπει να προσέξουμε τώρα ιδιαίτερα να εκπληρώσουμε τις υποσχέσεις που είχαμε δώσει. Δηλαδή, οι τροποποίησει του προϋπολισμού 2012 να μην συντρέχουν με τον προϋπολισμό 2013. Να γίνουν πολύ νωρίτερα, ώστε να μην υπάρξει ανάμειξη και έτσι να μπορούν να πληρωθούν ορισμένοι όροι. Είναι απαραίτητο λοιπόν η τροποποίηση του προϋπολογισμού για το 2012 να γίνει με τα ποσά που αναφέραμε και αυτό πριν από, τον, πριν από την θέσπιση του προϋπολογισμού του 2013. Κατά τα άλλα, οι συνάδελφοί μας γνωρίζουν ποιες είναι οι προτεραιότητές μας πρέπει οπωσδήποτε να είναι εγγυημένα τα κονδύλια για τα ευρωπαϊκά. δίκτυα. Το ίδιο ισχύει για τον Γαλιλαίο, για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Αυτά είναι τα προγράμματα για τα οποία χρειαζόμαστε απαραίτητα κονδύλια στον προπολογισμό. Επισημένω ωστόσο και πάλι κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα ότι είναι απαραίτητο να γίνουν οι διαπραγματεύσεις με σκληρό τρόπο και το Κοινοβούλιο πρέπει να λάβει σαφώς θέση. Διότι, όπως είπα, τα κονδύλια αυτά θα είναι πολύ σημαντικά και για τον προϋπολογισμό του 2014. Και δεν πρέπει να καταλήψουμε τις προτεραιότητες τις οποίες έχουμε ε, καθορίσει. Λίγα λόγια, αν επιτρέπετε από, την, από το επόμενα ως πρόεδρο, τονίζω και εγώ αυτά που είπαν ορισμένα μέλη μας για την θέσπιση προτεραιοτήτων στον, στον τομέα των μεταφορών για τη νέα στρατηγική του 2020. Είπαμε συχνά εδώ στην Επιτροπή μας ότι αν θέλει κανείς να δημιουργήσει ανάπτυξη, απασχόληση, αυτό, ε, το, οι μεταφορές είναι το ιδεώδες όχημα γι' αυτό. Με την κρίση, ωστόσο, η κρίση μάλλον έχει καταδείξει την ανάγκη να είμαστε πιο κριτικοί στον τομέα αυτό. Και βλέπω ότι όταν το Κοινοβούλιο έκανε τις διάφορες εκθέσεις στρατηγικής, οι μεταφορές κάπου βρίσκονταν σε τρεις-τέσσερις γραμμές σε μία από τις τελευταίες σελίδες. Τώρα το προφίλ των μεταφορών έχει ενισχυθεί, διότι hm, έχουν αναγνωρίσει όλοι και πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η συμβολή των μεταφορών και για την ανάπτυξη και για την απασχόληση, διότι δημιουργεί την υποδομή άλλωστε για πάρα πολλά χρόνια. Τα πρώτα χρόνια που ήμουν Ευρωβουλευτή είχα περάσει πολύ καιρό προσπαθώντα να πείσω τα άλλα μέλη τη Επιτροπή Προπολογισμών, τα μέλη μάλλον τη Επιτροπή Προπολογισμών, δεν, ε, η, η, η, πολιτική των μεταφορών είναι κάτι που χρειάζεται χρόνο. Δεν σημαίνει ότι εγκρίνονται τα κονδύλια σήμερα και δαπανώνται αύριο. Βέβαια δεν μπορεί να είναι και πάρα πάρα πολύ μακρές οι χρονικές περίοδοι. Οι προτεραιότητες αναφέρθηκαν επίσης. Το σύστημα σηματοδότησης των σιδηροδρόμων. Επίσης ο ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός. Είναι εδώ Υπάρχει βέβαια ένα κοινό υπόβαθρο που είναι το διαμεθοριακό στοιχείο. Αν μου πείτε ποια ήταν η μεγάλη αποτυχία των διευρωπαϊκών δικτύων στο παρελθόν, θα έλεγα ότι ήταν ένα ε, ε, σύνολο έργων τα οποία χαρακτηρίστηκαν από εθνικές προτιμήσεις. Χρειαζόμαστε ένα κόνσεπτ για τα διευρωπαϊκά δίκτυα που να είναι βασισμένο σε ευρωπαϊκές σε ευρωπαϊκό προβληματισμό, δηλαδή να υπάρχει μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για την οποία αναφέρθηκαν πολλοί βουλευτές πριν. Δεν με ενδιαφέρει να δοθούν χρήματα, να δοθούν κονδύλια για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα μέσα σε μια χώρα μέλος η οποία να μην προσφέρει ωστόσο συνολική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Θέλω έργα τα οποία να προσφέρουν ευρωπαϊκή θέμενη αξία. Και εδώ οι σιδηρόδρομοι είναι το κλασικό παράδειγμα. Βρισκόμαστε στο 2012 και δεν μπορούμε ακόμα ε, να επιτύχουμε τα τρένα να περάσουν από τα σύνορα. Είτε διότι το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι στη σωστή ε, συχνότητα ή στη σωστή ένταση ή διότι είναι διαφορετικές ε, το έβρος των τροχιών ή διότι τα σηματοδότηση είναι διαφορετική. Αυτές είναι οι ανοησίες που κάνουν οι εθνικές αρχές. Αυτός λοιπόν είναι ένας τομέας. Να δούμε λοιπόν από πού έχουμε ξεκινήσει. Θα σας βοηθήσουμε και στον ρόλο σας μέσα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για να βάλετε και εσείς στον προϋπολογισμό αυτές τις προτεραιότητες. Η τελευταία λέξη, για να βάλω και μια τρικλόποδιά αν μπορώ να πω έτσι, ένας λόγος που ποτέ δεν θα γίνω γενικός συγητής του προϋπολογισμού είναι διότι θα μπορούσα να κόψω πολλά κονδύλια περικόπτοντας την κοινή αγροτική πολιτική. Πριν πάθετε ωστόσο όλη η καρδιακή προσβολή σας, υπενθυμίζω ότι τα κονδύλια τη ΚΑΠ είναι τη τάξη των 40% του συνολικού προπολογισμού. και παρόλα αυτά δεν είναι προσανατολισμένη στις ανάγκες τη αγοράς. Εξακολουθεί να είναι βασισμένη σε μια μη αποδοτικότητα. Σύμφωνοι, τα θαύματα χρειάζονται κάπως περισσότερο χρόνο. Εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι δεν θα ζήσω για να το δω το θαύμα αυτό της βελτίωσης δηλαδή της αποδοτικότητας της ΚΑΠ. Κύριε Λαβή, έχετε πάλι το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η τελευταία σας αναφορά στην χρηματοδότηση της Γεωργίας με γαργαλά να πω κάποιες σκέψεις ε, αλλά τέλος πάντων δεν θα τα πω στην Επιτροπή Γεωργίας. Λοιπόν, προχωράω. Σας ευχαριστώ ε, προφανώς για τις διάφορες σκέψεις σας που με βοηθούν να κατανοήσω κάποιες ιδιαιτερότητες, κάποιες καταστάσεις και από την άλλη πλευρά μου επιτρέπουν αυτά που υπόθηκαν με τη σειρά μου να εκφράσω και εγώ κάποια πράγματα. Όπως είπατε και εσείς Πρόεδρε, στο τέλος της παρέμβασής σας οι μεταφορές είναι ένας από τους τομείς όπου έχει διαφορά μεταξύ, χρονική διαφορά μεταξύ αναλήψεως υποχρεώσεων και πληρωμών. Αυτή η διαφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε πάνω από 207 δισεκατομμύρια ε, ευρώ και το συνολικό ποσό των ποσών προς Και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους χρειάζεται, γίνεται αυτή η αίτηση για πληρωμών. Έχουν αληφθεί υποχρεώσεις για προγράμματα που χρηματοδοτούνται τα προηγούμενα χρόνια και αναπόφευτα λήγουν και θα πρέπει να πληρωθούν. Είναι σαφές ότι όσον αφορά αυτό το θέμα θα πρέπει σαν κοινοβούλιο ολόκληρο να υποστηρίξουμε το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ε, πληρωμές. Ελπίζουμε ότι στο πρόγραμμα προϋπολογισμού ε, το επόμενο να είναι αρκετά φιλόδοξη και ρεαλιστική όσον αφορά τις αναγκαίες, ε, τα αναγκαία χρήματα για να προχωρήσουν τα προγράμματα. Κατανοώ βεβαίως τις προτεραιότητές σας και είμαι σίγουρος ότι στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου και σε όλη τη διαδικασία του προπολογισμού θα μπορέσουμε να κινηθούμε και στο τέλος να έχουμε προπολογισμό που θα μπορεί να ευθυγραμμιστεί με τις προσδοκίες σας. Σωστά έλεγε ο συνάδελφος Μαρινέσκου ότι ο προπολογισμό του 2013 είναι ένα προπολογισμό παράξενο, διότι θα μπορούσε να είναι εκείνο του 2013, αλλά θα μπορούσε να είναι και ο προπολογισμό του 2014 ίσω. Διότι όπω όλοι παρατηρείτε τώρα, αν δεν καταλήξουν συμφωνία όσον αφορά το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, Κάτι που δυστυχώ πάντα υπάρχει σαν πιθανότητα. Ο προπολογισμό του 2013 θα γίνει προπολογισμό του 2014, διότι θα προσθεθεί απλώ ο πληθωρισμό, διότι αυτή είναι η συμφωνία μεταξύ των θεσμικών ε, οργάνων. Συμφωνία που έκαναν όταν εγκρίθηκε το προηγούμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάτι άλλο που αναφέρθηκε από πολλού συναδέλφου είναι το θέμα των, των πιλωτικών προγραμμάτων και των προπαρασκευαστικών δράσεων. Ε, για όλα αυτά Προφανώς ακολουθούμε τη διαδικασία του περσινού έτους όπως έλεγα, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα να γνωρίζουμε αν είναι εφαρμόσιμα αυτά ή τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το γνωρίζει. Αλλά σχετικό αριθμό και τους, πόρους που, τους οι που διατίθενται είναι γνωστοί όταν ξέρουμε τα περιθώρια που υπάρχουν εντός ε, των διαφόρων κονδυλίων, των διαφόρων γραμμών του προπολογισμού. Και το συνολικό περιβάλλον, όπω είπα, δεν είναι το καλύτερο δυνατόν η καταστάση όσον αφορά την καταβολή των πληρωμών. Ε, και είναι σε δύσκολη θέση αρκετά κράτη-μέλη λίγο τη οικονομική δυσκολία. Κάτι άλλο που ανέφεραν συνάδελφοι είναι η πολιτική του τουρισμού. Όπω ε, γνωρίζετε, είναι μια νέα αρμοδιότητα που δίνει η συνθήκη της Λισαβόνα, χωρίς όμως να δίνονται ειδικοί ε, πόροι στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και στη συνομιλίε συζητείται το θέμα. Από την άλλη πλευρά Έχουμε προφανώς κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες ήδη έχουν δρομολογηθεί στα πέστη των πιλωτικών προγραμμάτων και των προκατατικών δράσεων που θα μπορούσαμε όλα αυτά να τα υποστηρίξουμε. Αναφέρθηκε και σας ευχαριστώ, αναφέρθηκαν διάφορες προτεραιότητες όσον αφορά τα προγράμματα ε, Sky, Galileo κλπ, Μάρκο Πόλο, Σέζαρ, Διευρωπαϊκά Δίκτυα κλπ. Ε, θα προσπαθήσουμε για όλα αυτά ε, να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν στον προπολογισμό ε, και τι θα υπάρξει στον επόμενο προπολογισμό. Θα σας καλούσα σαν Επιτροπή να κάνετε αντικειμενικές αξιολογήσεις όσον αφορά τις δικές σας προτεραιότητες, όσον αφορά τα κονδύλια του προπολογισμού που σας ενδιαφέρουν στην Επιτροπή σας, αλλά να μας πείτε επίσης αν υπάρχουν και προτεραιότητες, διότι όλοι θέλουμε να προσθέσουμε περισσότερα, αλλά θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το γενικότερο πλαίσιο, που είναι ένα πλαίσιο δυσκολιών και κρίσης. Και ξέρουμε ότι δυστυχώς το Συμβούλιο πολύ συχνά στις συνομιλίες τελικές παρουσιάζεται και λέγοντας ότι το μέγιστο μπορώ να σας δώσω είναι μια αύξηση συν χ. Ήδη έχουμε επίσης κατευθείς γραμμές για τον προπολογισμό ότι δεν θα δεχτούμε τέτοιες προσεγγίσεις διότι και το Συμβούλιο θα πρέπει ενδεχομένως να υπομειστεί ευθύνε να πει που θέλει να κάνει τις περικοπές. Δεν μπορεί να αφήνει αυτή την καυτή πατάτα στα χέρια του Κοινοβουλίου όταν θα υπάρξουν πολιτικές που θα μπορέσουν να εφαρμοστούν λόγω ελλείψεως πόρων. Λοιπόν, το Συμβούλιο στην περίπτωση που θα θέλει να ακολουθήσει με τέτοια προσέγγιση θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να τονίσει ακριβώς και να δείξει που θέλει να κάνει συγκεκριμένες περικοπές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λαβία. Ε, εκτιμούμε το ότι ε, πάτε σε επιτροπές και ο η κυρία Μάιστρεν, η συγκήτρια για τον προπολογισμό μαζί με τους κοιόδης θα είναι σε συνεχή επαφή μαζί σας κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε στο επόμενο σημείο. Η, η γνωμοδότηση του κυρίου Μαρτσινκέβιτς για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και κατάρριση απόφασης 1364-2006. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, κύριε Μαρτσινκέβιτς. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, σημερινό αντικείμενο της συζήτησης ε, είναι οι διευρωπαϊκές ενεργειακές ε, υποδομές TEN-E. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τι βιωτικέ συνθήκε και την αποτελεσματικότητα των μεταφορών. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα ανεπτυγμένο διευρωπαϊκό σχέδιο, διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές που εξασφαλίζουν και οικονομική ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε αποφασιστικέ δράσει σε πλαίσια ανταγωνιστικότητες και ε, ανεφοδιασμού των ενεργειών. Φυσικά με συνέργεια μεταξύ ενεργειακών και μεταφορικών δικτύων. Χρειαζόμαστε εξυγχρονισμό ε, των ε, υποδομών στην Ευρώπη, όχι μόνο των ε, υποδομών μεταφορών, αλλά ταυτόχρονα και των ενεργειακών υποδομών. Στη γνωμοδότηση, η Επιτροπή Μεταφορών προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες προκειμένου να υλοποιήσουμε ε, τις, ε, τους στόχους αυτούς. Είχαμε την ανακοίνωση σχέση με το πολιτες δημοσιονομικο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, στο οποίο προτείνει τη δημιουργία της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη για την ολοκλήρωση των ε, υποδομών κατά προτεραιότητα ψηφιακών και ενεργειακών. Ε, στα πλαίσια αυτού του πλαισίου έχουμε 40 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ θα αφορούν την ενέργεια. Σε ό,τι αφορά το πεδίο αρμοδιότητας Επιτροπής ε, Μεταφορών, θα πρέπει να τονιστεί η χρησιμότητα της δημιουργίας συνεργειών κατά την υλοποίηση των ενέργων μεταφορικών υποδομών μέσω των ε, ενεργειακών υποδομών και το συντονισμό με τις μεταφορικές υποδομές, καθώς και την ευθυγράμμιση των διοικητικών διαδικασιών και των διαδικασιών που αφορούν τη χορήγηση αδειών και το περιβάλλον για τους κοινούς διαδρόμους ενέργειας και μεταφορών. Έχω πληροφορίες ε, που δείχνουν ότι είναι θετική η Ευρωπαϊκή Επιδρομή ως προς τις ε, αλλαγές αυτές, ε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα διοσυνοριακά και διακλαδικά προγράμματα, διατομιακά προγράμματα. Άλλα ζητήματα μεταφορών που αναφέρονται στη γνωμοδότηση αφορούν την μεταφορά πετρελαίου, αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας προς και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ιδιαίτερα για το πετρέλαιο και το αέριο χρησιμοποιούνται σιδηροδρομικές, ε, οδικές μεταφορές και, διαφορές, ε, και μεταφορές με πλοία. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση στις μεταφορές, ε, γιατί σε ό,τι αφορά τις μεταφορές θα πρέπει να επισημανούμε το 80% του εισαγόμενου αργού πετρελαίου μεταφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με δεξαμενόπλια. Ε, μάλιστα στις 15 ε, χώρες ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε προβλέπεται 7,8% αύξηση της, της κατανάλωσης του πετρελαίου μεταξύ 2010 και 2020. Γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε καλύτερες υποδομές μεταφοράς πετρελαίου με πετρελαγωγούς προκειμένου να εξασφαλίσουμε ασφάλεια εφοδιασμού και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Γιατί η μεταφορά πετρελαίων έχει σοβαρού περιβαλλοντικού κινδύνου. Σε περίπτωση διαταραχών του εφοδιασμού στο σύστημα στον αγωγό Ντρούσμπα, φιλία, οι περιορισμένε εναλλακτικέ δυνατότητε εφοδιασμού θα είχαν ω αποτέλεσμα σημαντική αύξηση τη κυκλοφορία των εξαεροπλοίων στην περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή τη Βαλτική, Μαύρη Θάλασσα και στα στενά του Βοσπόρου. Κάθε μήνα 3,5 με 5.000 πλοία διασχίζουν τα ύδατα τη Βαλτική θάλασσα. Περίπου 25% των πλοίων αυτών είναι δεξαμενόπλια και μεταφέρουν περίπου 170 εκατομμύρια τόνου πετρέλαιο ετησίω. Εκτός από μείωση του κινδύνου των μετραλοκυλίδων, η ελάττωση της κυκλοφορίας δεξαμενοπλοίων θα επέφερε επίσης μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και των εκπομπών οξιδίου του αζότου. Το φυσικό αέριο επίσης παίζει σημαντικό ρόλο για τις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ενέργειας, διότι αποτελεί βιώσιμη πηγή ενέργειας χαμηλών εκπομπών που εξασφαλίζει καθαρή ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Θα πρέπει λοιπόν ε, να, να κατά το δυνατόν η χρήση φυσικού αερίου. Επίσης ε, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στις μεταφορές. Έχουμε τις δύο δυνατότητες ε, φυσικού αερίου, υγροποιημένου και πεπιεσμένου φυσικού αερίου. Έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε και άμεσα στην υλοποίηση του στόχου των καθαρών μεταφορών. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές φυσικού αερίου, γι' αυτό και θα πρέπει να αναπτύξουμε τις υποδομές και να δημιουργήσουμε καλύτερες διασυνδέσεις και αγωγούς μεταξύ των χωρών μελών και επίσης ε, να προβλέψουμε και ε, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και επανεριοποίησης. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα σημεία και θα πρέπει να ενισχυθούν τα υφιστάμενα και να αναπτυχθούν νέα εθνικά δίκτυα μεταφορέ. Οι νέε κατευθυντήριε γραμμέ θα πρέπει επίση να καλύπτουν το ζήτημα των ενεργειακών νησίδων και τη απουσία διασυνδέσεων μεταξύ των εθνικών αγορών φυσικού αερίου, η οποία είναι αισθητή σε περιοχέ όπω η Βαλτική και η Κεντρική και η Ανατολική Ευρώπη. Έχω κάποιε προτάσει με βάση τα προαναφερθέντα. Για παράδειγμα, θα πρέπει να προαγάγουμε τι συνέργειε μεταξύ των εργών υποδομή Ευρωπαϊκή Ένωση, στους τομεί των μεταφορών και τη ενέργεια, μεταξύ άλλων μέσω τη ενθάρρυνση των αρμόδιων αρχών να χορηγούν κοινέ άδειε μεταξύ άλλων και στον τομέα περιβάλλοντο. Θα πρέπει περαιτέρω να αναπτύξουμε το υφιστάμενο δίκτυο αγωγών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να βελτιωθεί η σύνδεση μεταξύ των παλιών 12 και των νέων 15 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού με πετρέλαιο στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Θα πρέπει να μειωθεί ο δυνητικός κίνδυνος περιβαλλοντικών καταστροφών που προκαλώνται από την κυκλοφορία δεξαμενών Να προαγάγουμε το ρόλο των περιφερειακών τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου με ιδιαίτερη προσοχή στον ανεφοδιασμό των πλοίων στις σιδηροδρομικές μεταφορές και στι μεταφορές με φορτηγά να προαγάγουμε το ρόλο του φυσικού αερίου ως βιώσιμης πηγής ενέργειας, να επιδιώξουμε την ολοκλήρωση της αγοράς και να τερματίσουμε την απομόνωση των αγορών ενέργειας. Επίση θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημιουργία άρτιων και ευέλικτων εθνικών δικτύων μεταφοράς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την προσοχή και περιμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. κυρία Τσικάου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ως σκιώδης εισηγήτρια θα ήθελα να προβώ σε κάποια σχόλια σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει το ενεργειακό δίκτυο και το ηλεκτρικό δίκτυο να εξυγχρονιστεί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την αύξηση της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό είναι κάτι που θα αλλάξει το όλο σχήμα των δικτύων και του ενεργειακού μείγματος. Αυτό ισχύει και για το φυσικό αέριο. Αυξάνεται η ζήτηση. Το δίκτυο θα πρέπει να μπορεί να αντιδρά πιο γρήγορα. Θα πρέπει να αυξηθούν και οι δυνατότητες αποθήκευσης και να έχουμε περισσότερη προσφορά στον αφορά το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Ε, υπάρχει και μία μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δείχνει την ανάγκη ε, για επενδύσεις στην επόμενη περίοδο. Από τώρα μέχρι το 2020 χρειαζόμαστε περίπου 220 δισεκατομμύρια ευρώ για την ε, ανάπτυξη των μελλοντικών ενεργειακών δικτύων στην Ευρώπη. 140 από τα 220 δις θα πρέπει να διατεθούν για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως υψηλής τάσης. Ε, θα είναι υπόγεια, υποθαλάσσια δίκτυα, εναέρια, ε, αλλά χρειάζονται όμως να δοθούν χρήματα παρόλα αυτά. Ε, θα χρειαστούν στην Ευρώπη και δεκάδες δισεκατομμύρια ε, δίκτυα, εκατομμύρια για δίκτυα αφυσικού αερίου, υποποίηση και 25 δισεκατομμύρια περίπου για τη μείωση εκπομπών διεξουδίου του Ε, μεγάλα ποσά για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Περιμένουμε να αυξηθεί γενικά η ζήτηση ε, σημαντικά κατά την περίοδο, άρα χρειάζονται και επενδύσεις. Χρειάζεται μια νέα πολιτική. Μια πολιτική που να αποδεικνύει ότι υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών, να υπάρχει πραγματική εσωτερική αγορά που να μπορεί ε, να προμηθεύει και τι πιο απόμακρες περιοχές. Χρειάζεται να έχουμε και εναλλακτικά δίκτυα ενεργειακά ε, και θα πρέπει να εφαρμόζουμε μια πολιτική που θα επιτρέπει στις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας να ενταχθούν στα παραδοσιακά ενεργειακά δίκτυα. Θα ήθελα να πω ότι η πρόταση του κανονισμού προβλέπει και μια σειρά κανόνων για την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας θα πρέπει να έχουμε ε, σωστή ενεργειακή απόδοση, ε, να χρησιμοποιούμε περισσότερο εναλλακτικέ πηγέ ενέργεια και να υπάρχει και καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων ενεργειακών δικτύων. Αυτό ο κανονισμό σίγουρα θέτει προτεραιότητα για 12 διαδρόμου ε, και προγράμματα διάφορα σχετικά στρατηγικά στην Ευρώπη. Προβλέπει προδιαγραφέ για 7 κατηγορίες υποδομών κοινοφελών δικτύων ε, θα πρέπει να πούμε ότι προβλέπει και μέθοδο κανονισμός και διαδικασία που προβλέπει αρμονισμένη ανάλυση της σχέσης κόστους κόστους-οφέλους για τα διάφορα κοινοφελή προγράμματα όσον αφορά το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια. Προβλέπει επίσης κριτήρια επιλεξιμότητας για τα διάφορα προγράμματα που είναι κοινή τα προγράμματα τα οποία ε, υποστηρίζονται και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και σε επίπεδο μελετών και σε επίπεδο εκτελέσεως. Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης ότι από την πλευρά της Επιτροπής μας είναι σημαντικό να μπορούμε να ωφεληθούμε από μεταφορές οι οποίες ρηπαίνουν λιγότερο, δηλαδή ε, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ενεργειακές υποδομές που ρηπαίνουν λιγότερο. Θα σταματήσω για λίγο πάνω σε αυτό το θέμα. Οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια κανονικά χρησιμοποιούνται, ε, παράγονται σε τοπικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο και χρησιμοποιούνται εκεί. Αν πάρουμε όμω τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ε, και αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε πλήρω τη δυνατότητα που παρέχουν οι διάφοροι ε, ηλεκτρικοί φορεί, είναι σημαντικό να υπάρχει ισορροπία μεταξύ προστασίας ενεργείας, μεταφοράς ενεργείας κατανάλωσης ενέργειας ε, και της χρήσης ε, διαφόρων συστημάτων όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η, ο εύξηνο πόντο, η Μαύρη Θάλασσα έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μεταφορά της ενέργειας, κυρίως μεταφορά, για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Για να εγγυηθούμε την ασφαλή εφοδιασμό, εφοδιασμό συγγνώμη, τη Ευρωπαϊκή Ενώση Ενέργεια, χρειαζόμαστε μια πολιτική που θα έχει σαν στόχο τη μείωση τη εξάρτησή μα. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε νέου διαδρόμου εφοδιασμού οι ε, διάδρομοι νότια για το φυσικό αέριο είναι πάρα πολύ σημαντικοί για τον ασφαλή εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Βασική προτεραιότητα είναι ε, το πρόγραμμα Ναμπούκο, αλλά και άλλες προτεραιότητες έχουν σημασία. Όπως ο αγωγός φυσικού, η διάφορη αγωγή φυσικού αερίου, ο φυσικός αγωγός που θα ενώσει την Τουρκία με την Ιταλία και τη Ρουμανία με το Αζερμπαϊτζάν. Ε, και αυτή είναι διάδρομη πάρα πολύ σημαντική για τον ασφαλή εφοδιασμό της ε, Ευρωπαϊκής Ενώσης από την περιοχή Τευξίνου Πόντου. Θα πρέπει να αντιτικοποιήσουμε τη συνεργασία μας με τις χώρες ε, της περιοχής Τευξίνου Πόντου. Λοιπόν κύριε Πρόεδρε, είναι σημαντικό να αναπτύξουμε τις μεγάλες λιμενικές υποδομές, νέους τερματικούς σταθμούς στα λιμάνια, ούτως ώστε να περνά το υγροποιημένο φυσικό αέριο και να αποθηκεύεται το υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Γιατί διότι αυτό γίνεται όλο και πιο σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται επικοινομορφία στον αφορά τον εφοδιασμό και τις, ε, ε, τον τρόπο μεταφορών του φυσικού αερίου. Περιμένω να δω ποιε θα είναι οι τροπολογίε των συναδέλφων. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα συγχαρώ για μια ακόμη φορά τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω και δεν θέλω να πνίξω τη συζήτηση, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να συνομορφωθούμε το χρονοδιάγραμμα. Η κυρία Μάισνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να εξοικονομήσω λίγο χρόνο, αφού λέχθηκαν ήδη πολλά. Θα ευχαριστήσω πρώτον τον κύριο Ματσινκίεβιτς για την γνωμοδότησή του, η οποία συνδέεται με τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, με την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, αφού πρόκειται γενικά για υποδομές και ιδίως βέβαια των μεταφορών που απορροφούν και τα περισσότερα κονδύλια. Βέβαια και για την προμήθεια της ενέργειας και για της συχνότητα ευρώ Εδώ βρισκόμαστε βέβαια στην ενέργεια. Το ίδιο σημαντική υποδομή μεταφοράς της ενέργειας όπως και των μεταφορών. Γνωρίζω ότι σχεδιάζεται για παράδειγμα να χρησιμοποιηθεί η υποδομή των σιδηροδρόμων για τη μεταφορά των ενεργειών, της ενέργειας, συγγνώμη, ακόμη και της ολικής ενέργειας. Δεν είμαι βέβαια πώς μπορεί να γίνει αυτό, αλλά για παράδειγμα και από την θάλασσα πρόκειται να έρθει ενέργεια και η ενέργεια των αιωλικών πάρκων που χτίζονται και μέσα στη θάλασσα, πώς θα μεταφερθεί. Εκεί υπάρχουν και συνδυασμοί μεταξύ, δηλαδή θα μπορεί να γίνει ο συνδυασμός, η διασύνδεση μάλλον μεταξύ των υποδομών των μεταφορών και των υποδομών μεταφοράς ενέργειας. Είναι σημαντικό να αναζητήσουμε το, τις περισσότερες δυνατές συνέργειες, διότι ούτως ή άλλως αυτά θα κοστίσουν πολύ. Ας αποφευθεί λοιπόν με κάθε τρόπο η επικάλυψη. Διότι αυτό που θέλουμε είναι να υποστηριχθεί η ενιαία αγορά και με την υποδομή μεταφορών και με την υποδομή ενέργειας. Και μια ματιά τώρα πάλι στον προπολογισμό. Γι' αυτό και άλλωστε είπα ότι συνδέεται με την συζήτηση περί προϋπολογισμού και ιδίω τη διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη. Είναι σημαντικό να έχουμε τα κονδύλια στη διάθεσή μας διότι είναι λίγα τα χρήματα που ε, μπορούμε να διαθέτουμε για την ανάπτυξη της υποδομής. Τώρα, πιο συγκεκριμένα για τα όσα προτείνονται, δεν μπορώ να συμφωνήσω να περιορίσουμε ριζικά τη μεταφορά πετρελαίου με δεξαμενόπλια. Και βέβαια πρέπει να λάβουμε εκεί υπόψη κάποιε περιβαλλοντικέ επιβαρύνσει. Αν όμω δεν υπάρχουν άλλε εναλλακτικέ επιλογέ και εφόσον ούτω ή άλλω εξαρτώμεθα από το, από το πετρέλαιο, δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τα πετρελοφόρα, τα δεξαμενόπλια. Και ιδίω για τον Ντομινίκ Κρικέ που έχει αναλάβει την οδηγία για τα δεξαμενόπλια διπλού κήτου και θέλουμε να εξασφαλίσουμε νομοθετικά ότι τα δεξαμενόπλια θα είναι ασφαλέστερα. Σημαντικό επίσης είναι να ε, ελεγχθούν και οι αγωγοί, διότι πολλοί αγωγοί έχουν διαρροές και αυτό επιβαρύνει το περιβάλλον. Βέβαια δεν μπορούμε ξανά, λέω, να αφήσουμε τα δεξαμενόπλια. Τέλος, η υποδομή για μεταφορά του υγροποιημένου αερίου. Είναι μια εξαιρετική ενέργεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα καράβια. Υπάρχουν λιμάνια τα οποία φτιάχνουν από μόνα τους υποδομή για την αποθήκευση του υγροποιημένου αερίου. Αυτό είναι σημαντικό και για όλη την υποδομή της ενέργειας, διότι το υγροποιημένο αέριο δεν είναι δεδομένο μονάχα για τα πλοία, αλλά και για άλλα μέσα μεταφοράς. Γι' αυτό χαίρομαι λοιπόν που θα γίνουν προτάσεις και από τη δική μας πλευρά για το πώ μπορεί να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Ευχαριστώ. Ο κ. Κράμερ. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή για την έκθεση και βέβαια καλό είναι με αγωγούς να μπορούν να γίνονται μεταφορές αντί να γίνονται με δεξαμενόπλια. Αυτό δεν θα γίνει βέβαια σε όλες τις περιπτώσεις. Μπορεί όμως να γίνει εν μέρη διότι και ασφαλέστερο είναι και φιλικότερο προς το περιβάλλον. Άρα είναι καλό. Ποιος όμως θα πληρώσει. Έχουμε δύο τεράστιους αγωγούς, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο και δεν άκουσα να χρειάζονται αυτοί οι αγωγοί επιδοτήσεις. Μαλώνουν μάλιστα οι χώρε, όχι να περάσει από τη δική μου επικράτεια, όχι να περάσει από τη δική μου. Διότι πρόκειται η υπόθεση δισεκατομμυρίων. Το ερώτημα είναι, εάν κληθεί να, εάν είναι απαραίτητο να συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτέ τι χρηματοδοτήσει, ή αν μπορεί να τα κάνει ο κλάδο μόνο του. Από την ενέργεια κερδίζουν πολύ, πολλά λεφτά και υπάρχουν και περιθώρια επομένω. Παρ' όλα αυτά είναι χρήσιμο να γίνει και εδώ κάποια προσπάθεια συγκέντρωση όπου αυτό είναι απαραίτητο. Χωρί όμω να λησμονούμε την αποκεντρωμένη προμήθεια ενέργεια. Διότι η ενέργεια πρέπει να φτάσει παντού. Και στη Γερμανία, για παράδειγμα, τώρα μετά από την αλλαγή στην ενέργεια που καλωσόρισαν όλα τα κόμματα, τώρα έχει αρχίσει ο μεγάλος καυγάς. Μιλάμε μονάχα για τις μεγάλες επιφάνειες ε, απόκτησης ενέργειας, είτε για, τις, για ολικά πάρκα στις θάλασσες, είτε για την έρημο. Η δική μου θέση είναι τα μεγάλα μονοπόλια του ηλεκτρικού ρεύματος επιθυμούν να διατηρήσουν τα μονοπόλια τους και κυρίως την, την κεντρική τους θέση. Γι' αυτό και πρέπει να φροντίσουμε να είναι εξασφαλισμένη η αποκέντρωση. Για τα μεγάλα έργα το υγροποιημένο αέριο είναι τεχνολογία μετάβασης, διότι αυτό που θέλουμε είναι να είναι 100% ανανεώσιμη ενέργεια. Αν όμως θέλουμε να ξεφύγουμε από την πυρηνική ενέργεια και από τον ΑΚΑ θα χρειαστούμε το υγροποιημένο αέριο για κάποιο, για ε, χρονικό διάστημα. Και τέλος, όπως είπε και η κυρία Μάισνερ, πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω για τα πράγματα αυτά την σιδηροδρομική υποδομή, η οποία στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα πυκνή και όλοι οι αγωγοί που ζητούν τώρα να κατασκευαστούν οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να διασυνδεθούν με την υποδομή του σιδηροδρόμου. Το έχει προτείνει ήδη η Deutsche Bahn AG, η γερμανική σιδηρόδρομη. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο ότι δεν έχουμε τις απαραίτητες αυτές οδούς, αλλά υπάρχει κάποια αντίσταση διότι οι υποδομές είναι ευαίσθητες. Μπορεί να γίνει ως ο σιδηρόδρομος πρόδρομος και στις ε, νέες ενέργειες. Για παράδειγμα και με την χρήση της ενέργειας στα κτίρια του. Μπορούμε να κατευθύνουμε προς την, κίνηση, προς την κατεύθυνση αυτή ότι δηλαδή εδώ μπορεί να δημιουργηθεί μια συνεργασία μεταξύ των αγωγών και των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη. Να περνούν από τα ίδια σημεία, δηλαδή περνούν σιδηρόδρομοι. Ευχαριστώ, Ζέλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε πολύ καλή δράση στα πλαίσια του πολίτους δημοσιονομικού πλαισίου συμπυκνώνοντας διάφορες δράσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη. Βέβαια δεν είναι ακόμη ε, ιδεώδης η σύνδεση Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με Δυτική Ευρώπη. Μερικές φορές είναι καλύτερη η σύνδεσή μας με τρίτες χώρες, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. Γι' αυτό και συμφωνώ με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χαίρομαι και για την γνωμοδότηση του κυρίου Μαρτσινκέβιτς που επισήμανε ακριβώς αυτή τη διαφορά στις υποδομές μεταξύ των παλιών 15 και των νέων 12 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και αγωγή φυσικού αερίου που παραμένουν άδειοι. Και υπάρχει μερικές φορές πρόβλημα με την ενώ ταυτόχρονα υπάρχει πρόβλημα με τη μεταφορά του πετρελαίου. Γιατί να αφήνουμε άδειου του αγωγού ε, και να μεταφέρουμε το πετρέλαιο με σιδηροδρομικές ή ε, θαλάσσιες ε, μεταφορές. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερους πετρελαγωγούς, αν και ούτε και αυτή είναι η λύση για όλα μας τα προβλήματα. Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, χρειαζόμαστε σίγουρα τερματικούς σταθμούς για το υγροποιημένο αέριο και την εξασφάλιση καλύτερης διασύνδεσης μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας. Επίσης, θα πρέπει να απελευθερώσουμε την πρόσβαση στην αγορά και να διαφοροποιήσουμε την προμήθεια ενέργειας. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε ασφάλεια του ανεφοδιασμού. Η διαφοροποίηση είναι η λύση θα πρέπει να έχουμε διαφορετικούς ε, προμηθευτές. Χωρίς τέτοια διαφοροποίηση στην προμήθεια δεν πρόκειται να υλοποιήσουμε το στόχο της ασφάλειας του ενεργειακού ανεφοδιασμού. Ε, σε ό,τι αφορά τις κοινέ άδειε. Όταν μιλούμε για τον ηλεκτρισμό, Σίγουρα έχουμε χώρες που δεν συμμετέχουν στις περιφερειακές αγορές. Ούτε η Λιθουανία, ούτε η Λετωνία συμμετέχουν στις ε, ευρωπαϊκές χώρες. Ανήκουν στο δίκτυο της Ρωσίας. Αυτό είναι ένα, σημαντικό ζήτημα, μια πρόκληση που θα πρέπει να επιλύσουμε τα επόμενα χρόνια. Κύριε Συρικέ. Ε, λοιπόν, είναι ένα θέμα αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είμαι συνεισηγητή στον τομέα αυτό και εφόσον πρέπει να είμαι σύντομο, θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο προβλήματα τα οποία θεωρώ ότι διαβάζοντα την έκθεση αυτή και λαμβάνοντα υπόψη τη δουλειά που ήδη έγινε, ότι είναι σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, το θέμα το οποίο συζητάμε, η ενέργεια, είναι ζωτική σημασία. Χωρίς ενέργεια σταματούν τα πάντα. Δεν υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει δραστηριότητα, δεν υπάρχει ε, ζωή στο σπίτι. Όμως αυτό το θέμα αντιμετωπίζεται κάπως ε, σαν να μην είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάπως στο περιθώριο με το πρόσχημα ότι τελικά υπάρχουν πολλοί χρήματα γύρω από τα ενεργειακά προβλήματα και εφόσον υπάρχουν πολλά χρήματα του ιδιωτικού τομέα, δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με την αγορά η Ευρώπη. Στην πραγματικότητα υπάρχουν τεράστια προβλήματα χρηματοδότησης όσον αφορά το θέμα που αρέσει στον Πρόεδρο όσον αφορά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Στην πραγματικότητα ενδιαφέρεται η αγορά για πολλά τμήματα των μεταφορών, μεταφοράς ενέργειας, αλλά όχι για όλου του τομεί και κυρίω όσον αφορά τι διασυνδέσει στρατηγικέ ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. τη δυνατότητα να περάσουμε από ένα τύπο ενέργεια κλπ. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο μεγάλος μεταξύ διαφόρων ειδών ενέργεια. Μεγάλο είναι το πρόβλημα. Αντιλαμβανόμαστε από ό,τι είπαν οι παριστάμενοι ότι υπάρχει ε, πρόβλημα διασυνδέσεως μεταξύ χωρών, μεταξύ ειδών ενέργειας ε, όσον αφορά την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανταλλαγών, διότι δεν διαφέρει ε, την αγορά, ενδιαφέρει πολύ την αγορά. Υπάρχει ένα πρώτο πρόβλημα δηλαδή. Δηλαδή ότι η χρηματοδότηση των ενεργειακών δικτύων ε, είναι πάρα πολύ μεγάλη ορισμένα είδη ενέργεια και όχι για άλλα. Το βλέπουμε αυτό πάρα πολύ καλά, διότι στο Connecting ε, Europe Facilities, με τι επαφέ που είχαμε τα κράτη-μέλη, ποια ήταν η ιδέα του ότι δεν δίνουμε χρήματα για τα ενεργειακά δίκτυα. Πιθανότατα δεν δίνουμε χρήματα για τι διασυνέσει, για δυνατότητα χρήσεως ανανεωσίμων πηγών ενέργεια κλπ. Ε, και θα υπάρξουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. 250-260 δισεκατομμύρια χρειάζονται, εξαρτάται πώ θα το δούμε αλλά πού βρίσκονται στην ιδιωτική αγορά, η Ευρώπη και τα κάτι μέλη δεν θέλουν να δώσουν χρήματα και το αύριο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο νομίζω. Δεύτερο σχόλιο, πάντα μιλάμε για συνέργεια μεταξύ των δικτύων. Connecting Europe Facility λέμε είναι πάρα πολύ καλό, βάλουμε το broadcasting, την ενέργεια και τις μεταφορές στις ίδιες διατάξεις, διότι έτσι μπορούμε να έχουμε συνέργεια. Εγώ δεν βρίσκω τέτοιο πράγμα, λυπούμε. Δεν υπάρχει συνεργασία, πάρα πολύ λίγη. Υπάρχει κάποια συνέργεια όσον αφορά την παροχή ενεργείας, ε, όσον αφορά τα μέσα μεταφοράς και του μπαλίν, αλλά συνέργεια μεταξύ των δικτύων δεν υπάρχει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, με τα δίκτυα υψηλή τάση για τροφοδότηση των σιδηροδρομικών γραμμών, διότι αυτό δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά την ε, παροχή ε, Και το θέμα της τροφοδοσίας όσον αφορά τους πετρολογούς και τους αγωγούς φυσικού αερίου υπάρχει πρόβλημα ε, όσον αφορά τα ατυχήματα κλπ. θα έχουμε τεράστια προβλήματα χρηματοδότηση, όπω σα είπα, όσον αφορά τι ενεργειακέ υποδομέ διανομή ενέργεια, διανομή ενέργεια που θα δίνει η ευρωπαϊκή προστιθέμενη ε, αξία και θα πρέπει να εργαστούμε πάρα πολύ ώστε να πετύχουμε τη συνέργεια που θέλουμε να πετύχουμε. Ο κύριο Κούν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καθώ επίση και τον εισηγητή κύριο Μάτσιν Κίβιτς. Δεν πρόκειται απλά για συζήτηση για το πώ μπορούμε να βελτιώσουμε τι υποδομέ στην Ευρώπη, είναι περισσότερο συζήτηση στρατηγικής. Και όταν συζητούμε πώς θα στερεωθεί η θέση της Ευρώπης στον ανταγωνισμό παγκόσμια, όταν βλέπουμε τι κάνουν οι Αμερικανοί, τι κάνουν οι Ασιάτες, πρέπει να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο στις σκέψεις μας. Και είναι απαραίτητο να δώσουμε καθαρά τις κατευθυντήριες γραμμές για την εξασφάλιση προμήθειας της ενέργειας στην Ευρώπη. Ασφαλώς πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αλλά ασφαλώς και άνθρακα και ανανεώσιμες ενέργειες που θα παίξουν πολύ κεντρικό ρόλο. Αυτή η υποδομή που είναι απαραίτητη ώστε από εκεί που παράγεται ενέργεια να φτάνει μέχρι εκεί που καταναλώνεται. Αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολήσει τώρα και βέβαια και το ερώτημα πώς θα συνοδεύσουν, πώς θα παρακολουθήσουν τις πολιτικές αυτές οι πολίτες μας. Αυτά όλα πρέπει να ανέβουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Αυτό θέλω να πω. Έχουν σχέση με την υποδομή των μεταφορών και τον αυτοκινητόδρομο και τον σιδηρόδρομο και το αεροπλάνο και το πλοίο που αυτά είναι ημίς του σώματος της Ευρώπης ενώ η ενέργεια είναι το αίμα. Και αυτά είναι που απαιτούν και οι πολίτες από εμάς τους υπεύθυνου πολιτικούς. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η συζήτηση. Κατά πόσο δηλαδή αυτή η κρίσιμη υποδομή θα πρέπει να παραμείνει στα χέρια του δημοσίου, να μην ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα. Κρίσιμη υποδομή. Ανταγωνισμός να υπάρχει. Αλλά οι κρίσιμες βιομηχανίες η αγωγή. Εκεί πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ καλά κατά πόσον θα διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μας. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν τώρα, ο κ. Μόμο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημαντική αυτή συζήτηση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Μαρτινκίεβιτς, τον εισηγητή, για την έξοχη γνωμοδότησή του και τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά στη συζήτηση και στη διατύπωση του κειμένου. Ακούγοντας συζήτηση διαβάζοντας την έκθεση, την γνωμοδότηση μάλλον, πρέπει να πω ότι βλέπω ότι υπάρχει εντύπωση ότι συμφωνούμε επί των βασικών σημείων. Όταν κάναμε την πρότασή μας, στόχος βασικός ήταν η διασύνδεση μεταξύ των αγορών, επιτρέποντας τη χρήση ανανεωσίμων πηγών ενέργειας, περισσότερες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Ευρώπη. Είχαμε στατηγικούς στόχους υπόψη μας, αλλάζοντας τα ενεργειακά συστήματα. Θέλουμε να δούμε πώς πρέπει να είναι στο μέλλον και πώς μπορεί να είναι στο μέλλον ανταγωνιστική Ευρώπη, πώς μπορεί να αλλάξουμε τα συστήματα, με λόγια. Οπότε ακολουθούμε παρόμοιες γραμμές και χαίρομαι πολύ που ακούω αυτά που λέει το Κοινοβούλιο και ότι προσεγγίζει το θέμα παρομοίως. Αυτό που θέλω να τονίσω και είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι χρειάζονται συνέργειες μεταξύ διαφόρων τομέων και, και γι' αυτό, όπως ίσως γνωρίζετε, έχουμε προτείνει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, αυτές που συζητούμε σήμερα. Και για τις μεταφορές και για τις υποδομές της πληροφορικής. Όλα αυτά συναθρίζονται σε μία πρόταση με το μέσο για, την, ε, να ενώσουμε την Ευρώπη, Connecting Europe Facility. Θέλουμε να δούμε πώς υπάρχουν διαδράσεις μεταξύ των διαφόρων υποδομών. Και γιατί πρέπει να εκμεταλλευτούμε συνέργειες και πώς. Βλέπουμε στην πρόταση ότι προτείνουμε περισσότερη σηματοδότηση για πιο δύσκολα προγράμματα και τα πλούστερα ε, προγράμματα είναι αυτά που συνδυάζουν διάφορους τομείς. Προσπαθούμε να το λάβουμε υπόψη. Και αν δείτε τις κατευθύντες γραμμές και το Connecting Europe Facility σαν κοινή πρόταση, τότε η εικόνα γίνεται σαφέστερη. Και κάτι επιπλέον. Όσον αφορά το πετρέλαιο και την ανάγκη συνδέσεως υποδομών Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό. Χρειαζόμαστε καλύτερες διασυνδέσεις για τα δηληστήρια που επεξεργάζουν το πετρέλαιο. Θέλουμε λοιπόν τις υποδομές πετρελαίου να τις έχουμε στις κατευθυντικές γραμμές. Πιο σημαντικό είναι η ασφάλεια εφοδια... ασφαλής που συνδέεται με το θέμα της διασύνδεσης. Το θέμα των δηληστηρίων αφορά περισσότερο τα κράτη-μέλη. Αλλά όσον αυτό το πετρέλαιο, ίσω έχουμε μία πηγή. Τα κράτη-μέλη εξαρτώνται από μία μοναδική πηγή για το πετρέλαιο. Πώ θα καλυφθεί το κόστο των υποδομών. Για το πετρέλαιο μπορεί να θεωρηθούν κοινοφελεί υπηρεσίε. Μπορεί να επιταχυνθεί η αδειοδότηση. δεν προτείνεται συγκεκριμένη χρηματοδότηση για τη σύνδεση, διότι μιλάμε κυρίως για ιδιωτικές υποδομές, δεν ρυθμίζονται και δεν είναι ανοιχτέ ε, σε όλους την αγορά και διαφέρει το πετρέλαιο από ότι ο ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, οι υποδομές τους. Ε, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Ελπίζω η πρότασή μας να προχωρήσει ε, χωρίς να αλλάξει πολύ η μορφή της. Ευχαριστώ. Κύριε... Θέλετε να προσθέσετε κάτι κύριε Μαρτσικέβιτς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα σχόλια των συναδέλφων. Θα ήθελα να πω καταρχήν, μιλούμε για τις κατευθυντήριες γραμμές ό,τι αφορά τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα και μιλούμε για την επόμενη ε, για τις επόμενες προοπτικές 2014-2020, στη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή πολιτική της κάθε χώρας, θα ήθελα να πω ότι η κάθε χώρα έχει τη δική της ενεργειακή πολιτική και το δικό της ενεργειακό μείγμα που το δημιουργεί, ανάλογα με τις ανάγκες και τους σκοπούς. Και βέβαια κάθε χώρα σε διαφορετικό βαθμό υλοποιεί τους ενεργειακούς της στόχους. Και φυσικά δεν μπορούμε τεχνητά να τα ενοποιήσουμε όλα. Θα πρέπει να έρθει μια πιο φυσιολογική διαδικασία. Σε ό,τι αφορά την μεταφορά ενέργειας με σιδηροδρόμους. Νομίζω ότι είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Γίνονται μεταφορές ε, βουτανίου, για παράδειγμα, με σιδηροδρομικές ε, μεταφορές, με σιδηροδρόμους. Και υπάρχει δυνατότητα τέτοιες μεταφορές, όπως και με τις οδικές μεταφορές. Ό,τι αφορά τις, ε, είναι, ε, τις ε, νομίζω ότι είναι εύκολο να, εύκολο να δημιουργηθεί διασύνδεση συνδέοντας τους αγωγούς με τις ε, μεταφορές. Σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές ε, ανησυχίες και το θέμα αυτό είναι σημαντικό. Έχουμε και, διαφορετικές περιβαλλον... Έχουμε περιβαλλοντικές και προσπαθούμε να μεταφέρουμε την ενέργεια με διαφορετικές ε, περιβαλλοντικές ανησυχίες. Για παράδειγμα, βλέπουμε την νέα πολιτική των, ε, της ε, Γερμανίας που αποφάσισε να σταματήσει την χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα. Διαφορετικές είναι και εδώ οι πολιτικές. Επίσης, οι διάφορες χώρες επενδύουν με διαφορετικό τρόπο στους φορείς της ενέργειας. Βλέπουμε και τους εταίρους μας στην Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Ινδία. Θα πρέπει ταυτόχρονα, λαμβάνοντα υπόψη τι περιβαλλοντικέ μα ανησυχίε, να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητά μα και να διαμορφώσουμε και το δικό μα ενεργειακό μείγμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφου ε, για τι ε, πολύ χρήσιμε παρατηρήσει του. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ακούσαμε. Πάντως, ε, σε συνεργασία με τους σκιώδεις ηγητές, θα διαμορφώσουμε μια συνενετική γνωμοδότηση που πιστεύω θα είναι ικανοποιητική για την Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Μασινκίεβιτς, Μασινκίεβιτς συγγνώμη. The 29 e e. Απριλίου είναι η προθεσμία κατάθεση των τροπολογιών. Α, όχι, διορθώνει ο 11 Απριλίου, ζητούμε συγγνώμη. Και τελευταίο θέμα, η έκθεση του κυρίου Κόλιτσεκ για την συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερικής Ανάπτυξης στην επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Έχει αμέσως τον λόγο γιατί περιμένει αρκετή ώρα. Και έχω ήδη εγγεγραμμένους ε, τέσσερις ε, συναδέλφους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μου χρειαστεί μισή ώρα, εγώ προσωπικά δηλαδή. Θα, συνεχίσω να μιλώ τσεχικά βέβαια τώρα, αν μου επιτρέπετε. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για δίκτυα και για μεγάλες, μεγάλες πολιτικές η έκθεση που έχω συντάξει, η γνωμοδότησή μου, αναφέρεται σε ελάσσονα περιφερειακά προγράμματα συνεργασίας που είναι επίσης πολύ σημαντικά και είναι σημαντικά και για τα μεγάλα δίκτυα διότι στοχεύουν να διασφαλίσουν διαμεθοριακές διασυνδέσεις για μικρότερα έργα, ε, στο ποδηλατοδρόμους, ε, στο ε, επικοινωνίες διαμεθοριακά κλπ. που όμως είναι σημαντικά για τους ανθρώπους που κατοικούν στις περιοχές αυτές. Διότι χωρίς αυτά δεν θα είχε νόημα να συζητούνται άλλα θέματα όπως αυτά του κύριου Μαρτσινκιέβιτ. Με άλλα λόγια, πρέπει να τονώσουμε την διαπεριφερειακή συνεργασία όπως, την έχουμε, δει και στο, όπως έχουμε δει στο παρελθόν άλλωστε και νομίζω επίσης ότι πρέπει να ε, ρίξουμε, δώσουμε περισσότερη έμφαση στα αποτελέσματα, να μειώσουμε το γραφειοκρατικό κόστος, κάτι το οποίο βέβαια οφείλει να γίνει παντού και κυρίως, αυτό πρέπει να τονιστεί, να απαιτούμε πάντοτε το Συμβούλιο να μας υποβάλει εκθέσεις για την πραγματική αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών. Δεν είναι δυνατόν να ασκείται μια πολιτική επί μια επταετία χωρίς καμία παρέμβαση, χωρίς κανείς να έχει μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της. Η πρόταση επίσης προβλέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος σε ορισμένα θέματα. Προσωπικά τονίζω την διασύνδεση μεταφορών και τουρισμού και αν εξετάσετε ορισμένε από τις τροπολογίες που έχουμε μπροστά μας βλέπετε να μιλούν για διασυνδέσεις διαμεθοριακές για ορισμένες από τις βιομηχανίες οι οποίες γνώρισαν μια σημαντική παρακμή είναι πράγματα τα οποία τα συζητούμε ήδη εδώ και μια οκταετία περίπου και τα θέματα αυτά ε, είναι τομέων που έχουν ανάγκη από στήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών. Το ίδιο χρειάζεται στήριξη η περαιτέρω ανάπτυξη της υποδομής γιατί σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις περιοχές αυτές επίσης και μικρές επιχειρήσεις που ωστόσο είναι πολύ σημαντικές για την εξασφάλιση της απασχόλησης. Το ίδιο είναι σημαντικό να γίνει προσπάθεια το επίπεδο, το βιωτικό επίπεδο να παραμείνει σε συγκρίσιμα επίπεδα με αυτά των πιο αναπτυγμένων περιοχών. Θα ήθελα επίσης να συμφωνήσετε να συζητήσουμε ορισμένα από τα θέματα που, είχαμε, που έχουμε ήδη συζητήσει στην Επιτροπή μας, ε, κάποιες συνέργειες μεταξύ της γεωργίας και της περιφερειακής συνεργασίας με στόχο ιδιαίτερα την βελτίωση των υποδομών. Όπως είπα, είτε πρόκειται για δρόμους, είτε πρόκειται για τον αγροτοτουρισμό, πράγματα δηλαδή τα οποία θα βελτιώσουν το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων των περιοχών αυτών. Βελτίωση δηλαδή των συνθήκων στις περιφέρειες αυτές προώθηση της συνεργασίας. Υπάρχουν ορισμένα έργα στα τσεχοβαβαρικά σύνορα, ορισμένα σχέδια δηλαδή, τα οποία ορισμένα από αυτά είναι δυνατόν να υλοποιηθούν και νομίζω το πρόγραμμά μας μπορεί να βασιστεί σε αυτά τα ήδη φυστάμενα σχέδια. Ευχαριστώ αυτά από τη δική μου πλευρά και Αναμένω τώρα τα σχόλιά σας, τα οποία θα περάσω μετά και σε άλλες επιτροπές. Γιος Φιδάντσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αντικαθιστώ τον συνάδελφο Ταταρέλα που είναι πραγματικό σκιώδη όσον αφορά αυτή την έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Είναι πολύ ουσιαστική η δουλειά, πέντε τροπολογίε, αλλά αφορούν ε, την ουσία του θέματος θετική τοποθέτηση όσον αφορά τις πέντε τροπολογίες, βέβαια κυρίως όσον αφορά τις τροπολογίες που αφορούν την διασυνοριακή συνεργασία, όσον αφορά τα ειδικά θέματα της διασύνδεσης των ε, μεταφορών και τη σχέση με την πολιτική του τουρισμού συμφωνούμε επίσης και με την πρόβλεψη εκθέσεων πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου Περιοδική Εκθέσεων αφορά την αποτελεσματικότητα των μέσων για την πολιτική συνοχή. Θα, στη φάση των τροπολογιών θα θεωρούσαμε θα, θα πρέπει να απευθύνουμε έκκληση όσον αφορά το διασυνοριακό τουρισμού, να αναφέρεται όχι μόνο σε τελογικές σκέψεις όπως προβλέπεται για την ώρα από τον εισηγητή αλλά να αναφέρεται και στο διατακτικό του κειμένου, στο κείμενο του κανονισμού Πιστεύουμε επίσης ότι θα ήταν καλό να πιέσουμε περισσότερο για το συντονισμό που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των διαφόρων ταμείων για περιφερειακή ανάπτυξη και το, ΦΕΖ, και το Αγροτικό Ταμείο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και για το Ταμείο για την Αλία και τις ε, πολιτικές για τη θάλασσα και να δοηθεί ιδιαίτερη σημασία στις ευρωπαϊκές ομάδες εδαφικού συντονισμού που είναι νέες μορφές διασυνοριακής συνεργασίας και στις περιφέρειες που ξεκίνησαν να εφαρμόζουν αυτή την προσέγγιση άρχισαν να παράγονται καλά αποτελέσματα. Από ό,τι κατάλαβα και η Επιτροπή Ρέτζη και η, που είναι Επιτροπή Καθήλια και η Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή ε, θα υποβάλουν ειδικέ ε, τροπολογίες. Ελπίζουμε που δεν θα επεξεργάζονται εξ αρχή στην πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι είναι σωστή προσέγγιση του συγητού να επικεντρωθούμε επί λίγων συγκεκριμένων σημείων όσον αφορά τι ε, τροπολογίε. Ο κύριος Λιμπεράτσκι για τους σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή, τον κύριο Γιώργο Μυρκοχλίτσεκ, για την γνωμοδότησή του θα ήθελα να επικεντρωθώ στα εξή. Καταρχήν, το σχέδιο γνωμοδότησης ε, ε, ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της πολιτικής μας ομάδας που ήθελε μια στρατηγική, ένα στρατηγικό συντονισμό και στρατηγικές κατευθυντήρες γραμμές για τα προγράμματα διασυνοριακής ε, εδαφικής συνεργασίας. Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να έχουμε επίγνωση ότι εμείς με την γνωμοδότηση αυτή δεν έχουμε σημαντικά χρηματοδοτικά μέσα. Θα πρέπει να βρούμε διαφορετικό τρόπο διαχείρισης με τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά μέσα, γιατί συμπληρωματικά δεν πρόκειται να έχουμε κονδύλια. Στο σημείο 4, σε ό,τι αφορά την ε, επιρροή μας στον προϋπολογισμό και το κονδύλιο του Ταμείου Συνοχής. Είναι αντίστοιχο το κονδύλιο με αυτό που είχαμε στην ε, περίοδο 2007-2013. Οπότε το σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε νέα ε, χρηματοδοτικά μέσα, δεν έχουμε νέα κονδύλια, αλλά διαφορετική κατανομή των υφιστάμενων κονδυλίων. Χρειαζόμαστε περισσότερη διασυνοριακή συνεργασία, διακρατική συνεργασία και διαπεριφερειακή συνεργασία. Πρόκειται για τρεις κατηγορίες συνεργασίας που αναφέρονται και θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε επιλεκτικούς ε, ε, διακρατικούς στόχους και θεματικούς στόχους. Μόνο έτσι με ιεράξη των προτεραιοτήτων θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Βέβαια δεν είναι αντίστοιχος ο ενθουσιασμός πολλές φορές ε, των κρατών μελών. Γιατί, όπως αναφέρεται στο σημείο 21, έχουμε, θα πρέπει να δούμε τη διαφορά μεταξύ των δικαιούχων, των βασικών δικαιούχων και να μην αυξήσουμε ε, την εθνική συγχρηματοδότηση, αλλά να, αυξηθεί, ε, να ενισχυθεί ο ρόλος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να δούμε τη σχέση μεταξύ του πεδίου και του στόχου. Αναφέρεται στο 27 πρώτο εδάφιο. Δηλαδή να αναφερθούν τα διακρατικά, διασυνοριακά ε, τα προγράμματα συνεργασίας και κατηγορίες παρέμβασης. Θα ήθελα αυτά τα σημεία ε, να τα λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ξεκινήσει διαβουλεύσεις και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να μην έχει μόνο διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες, όπως έγινε για το σχέδιο κανονισμού. Γιατί σε τελική ανάλυση εμείς δεν ξέρουμε ποιοι ήταν οι συμβουλάτορες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ποιους έγιναν οι διαβουλεύσεις. Θέλουμε έναν κανονισμό να είναι, που θα είναι πλήρης, μεστός, δηλαδή να αναφέρεται και στον προγραμματισμό και στην ε, παρακολούθηση, στον έλεγχο, στη διαχείριση, στη διαπίστευση και στον έλεγχο της πιστοποίησης. Θα πρέπει ε, να είναι πλήρης με όλα αυτά τα σημεία ο κανονισμός. Επίσης, ε, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν υπόψη ότι τα κονδύλια που είχαν θα αλλάξουν κάπως, αλλά ο ίδιος ο κανονισμός δεν θα πρέπει να αντιτάσσεται στους ε, στόχους μας. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για την γνωμοδότησή του και σας διαβεβαιώνω για την προθυμία της ε, συνεργασίας και υποστήριξης ε, μέσω και των τροπολογιών που θα καταθέσουμε. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Liberaski. Κύριε Ρούγγιας, θα ήθελα να καλωσορίσω τώρα την ομάδα επισκεπτών της κυρίας Φώστερ από το Πόιντον, βόρειο-δυτική ε, Αγγλία. Ξέρετε ότι η Βορειοδυτική Αγγλία είναι η καταπληκτικότερη περιοχή, η καταπληκτικότερη περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Επαναλαμβάνω, η ομάδα επισκεπτών είναι προσκεκλημένη της κυρίας Φώστερ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή ε, Μεταφορών και Τουρισμού, κύριος Ούτζιας, για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα ασχολούμαστε με ένα θέμα από διαφορετική οπτική γωνία από αυτή που έχουμε συνηθίσει. Μιλάμε πάντα για μεγάλα δίκτυα, μιλάμε για μεγάλες διασυνδέσεις. Σκεφτόμαστε μεγάλη κλίμακα, όμως σήμερα οδηγούμεθα να τα βλέπουμε σε πιο μικρή κλίμακα. Θέλουμε εδαφική συνεργασία, να την προωθήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξέρουμε, υιοθέτησε μια ανακοίνωση όσον αφορά ε, σε σχέση με την ε, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Υπογραμμίζεται η σημασία που έχει η συνεργασία η διασυνοριακή. Έχω κα... να εκφράσω δύο σκέψεις γενικές όσον αφορά τον κανονισμό. Πρώτον, πρέπει να υποστηρίξουμε κάποιες γραμμές που διαφάνησαν ήδη στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πιο σημαντική γραμμή είναι ότι θα πρέπει να θέσουμε τροχοπέδι στο περιεχόμενο της ανακοίνωσης, όπου εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πράξη ε, παίρνει κάποια προνόμια που θα έπρεπε να διατηρηθούν στον πραγματισμό του Κοινοβουλίου, κυρίως όσον αφορά την εξουσία τη δυνατότητα να αθετούνται οι κατεξουσιοδότηση πράξεις. Εν αυτή τη ενία είναι θετική η τροπολογία που υπευλήθη από πλευρά εισηγητού του κυρίου Κολίτσεκ. Τον ευχαριστώ πολύ για την καλή δουλειά που έκανε. Που ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή να περιοριστεί αυτή η εξουσία. Δεύτερη πτυχή που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η εξή. Πώς περιγράφεται το πλαίσιο της governance, δηλαδή σε επίπεδο προγραμματισμού, γενικού προγραμματισμού, πρέπει να υπάρχει διασύνδεση με τον προγραμματισμό των περιφερειών. Και αυτή είναι η άλλη σημαντική πτυχή, πιστεύω, που θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα και να δώσουμε σημασία. Γι' αυτό ο περιορισμός των προτεραιοτήτων του κειμένου θα πρέπει να περιέχει δηλαδή, το κείμενο το πολύ τέσσερι προτεραιότητε. Και θα πρέπει να δούμε διασυνδέσεις μεταξύ διασυνοριακών προτεραιοτήτων, ούτω ώστε να μην υπάρχει διάχυση στόχων. Όπως είδαμε από την έκθεση για τη λειτουργία των προγραμμάτων Interreg του 2000, από το 2000 μέχρι 2006. Θέλουμε καλύτερο καθορισμό των προτεραιοτήτων, ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διασύνδεση μεταξύ διαφόρων προγραμμάτων και έτσι μπορούμε να πετυχαίνουμε καλύτερους στόχους. Θα πρέπει να θέσουμε εγώ το στόχο πιστεύω, δηλαδή να εντοπίσουμε προτεραιότητες ακριβεί και να μπορέσουμε ε, στο τέλος διαδρομής του προγραμματισμού να βλέπουμε την επίτευξη των στόχων. Μείωση του, της πατάλης, ε, μείωση ε, των στόχων ε, και καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή πρέπει να είναι η στόχη του κανονισμού. Και κάτι που ήδη υπόθηκε, αλλά πιστεύω ότι ποτέ δεν αρκεί να το επαναλαμβάνουμε. Ο διεθνής τουρισμός, δηλαδή πώς μπορούμε να τον προωθήσουμε όπως έλεγε και πριν ο συνάδελφος Φιντάνσα. Θέλουμε αυτό να αναφέρεται όχι σε αιτιολογική σκέψη, αλλά σε συγκεκριμένες προτάσεις. Να δώσουν προτεραιότητες στις περιοχές αυτές που έχουν ως σημαντική πηγή της ανάπτυξής τους τον τουρισμό. Thank you very much, Mr. Kramer. Ευχαριστώ, Κράμερ, των Πράσινων. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή κ. Κόλιτσεκ για την δουλειά του που έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις διαμεθοριακές μεταφορικές, μεταφορές ή συγκοινωνίες. Γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κινούνται παραπάνω από μια, σε μια ακτίνα από παραπάνω από 50 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικία. Πρόκειται για μια πραγματικότητα. Απ' την άλλη μεριά δεν βρίσκει απήχηση στην οικονομική, δημοσιονομική πραγματικότητα. Άρα χρειάζεται βελτίωση. Αν δείτε τον χάρτη μεταφορών Τη Ευρώπη θα δείτε να μην έχει ανάξει τίποτα τα τελευταία 20 χρόνια. Τα κενά που επισημιώνονταν τότε εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα και συμπίπτουν με τα σύνορα. Άρα δεν καταφέραμε να συνδέσουμε την Ευρώπη. Και εδώ βέβαια το ρόλο πρέπει να αναλάβουν οι περιφέρειες, διότι με τον τρόπο αυτό θα έρθουν πιο κοντά, θα γνωριστούν κλπ. Θα σας πω λίγα παραδείγματα. Το 1972 μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας υπήρχαν ακόμα 18 σιδηροδρομικές συνδέσεις την ημέρα. Μετά, τώρα 23, 23 χρόνια μετά από την πτώση του στίχους, θα λέγατε ότι υπάρχουν 50. Όχι. Υπάρχουν 10 μόνο. Το Βερολίνο, Μπρέσλαου. Χρειαζόμασταν το 1980 για τα 800 χιλιόμετρα 6 ώρες. Σήμερα από τη γερμανική πλευρά, από το Βερολίνο μέχρι το Κότμπους, κάναμε ηλεκτροκίνηση της γραμμής Επίσης, οι Πολωνοί από τη δική τους μεριά, το μεγαλύτερο μέρος, λείπει ηλεκτροκίνηση. Δεν κάνουν τίποτα για 50 χιλιόμετρα, 50 χιλιόμετρα κενό της ηλεκτροκίνησης. Από την άλλη μεριά έχουν δώσει δισεκατομμύρια για το αεροδρόμιο της Στουτγάρδης, για διάφορες σύραγγες, για τα αυτοκίνητα κτλ. Και δεν δίνουν τα χρήματα αυτά για το 50 χιλιόμετρα. Τώρα, Βερολίνο-Στετίνο 30 χιλιόμετρα ηλεκτροκίνηση, 5 χιλιόμετρα από πολωνικής πλευρά, 25 από γερμανική. Οι Πολωνοί λένε ότι εμεί θα φτιάξουμε τα 5 χιλιόμετρα, όταν πρώτοι οι Γερμανοί θα φτιάξουν τα 25 χιλιόμετρα. Μετά από την εμπειρία που έχουν με το Βερολίνο Μπρέσλαο, του καταλαβαίνω του Πολωνούς, δίκιο έχουν. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποια κίνητρα, κάποιε πρωτοβουλίε που ε, να προχωρήσουν τα πράγματα αυτά. Θα σα μπορούσα να σα πω και πολλά άλλα παραδείγματα, αλλά θα περιοριστώ μόνο σε αυτά. Για την υποδομή των μεταφορών, τα είπατε και άλλες φορές, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μοναχά τους δρόμους. Θα ήθελα να περιλάβετε τη λέξη βιώσιμος, που τη δυστυχώς σήμερα στην ψηφοφορία. Πρέπει να είναι λοιπόν βιώσιμες οι μεταφορές αυτές. Ο δε τουρισμός έχει εδώ ιδιαίτερη συνάφεια και είναι σωστό που αναφέρεται. Μπορεί όμως να τονωθεί περισσότερο ο τουρισμός, μπορεί να τονιστεί ο ρόλος του, διότι γνωρίζουμε ότι ο πολλή τουρισμός μπορεί να καταστρέψει εν τέλει τον τουρισμό. Χρειαζόμαστε και έχουμε μια τάση στην Ευρώπη προς τον οικολογικό τουρισμό. Κάθε χρόνο αυξάνονται 20% οι ποδηλάτες που κάνουν τουρισμό. Και όλες οι μελέτες τα λένε, ένα θαυμάσιο φυλάδιο υπάρχει εκεί μπροστά, ότι οι ποδηλάτε δαπανούν και περισσότερα από του αυτοκινητιστέ όταν κινούνται για τουρισμό. μπορούν και από τις δύο πλευρές των συνόρων ε, έχουν θαυμάσιες ε, έχουν θαυμάσιες ε, περιοχές, θαυμάσιες τοποθεσίες και πολλές περιοχές μπορούν να διασυνδεθούν. Σλοβακία, Αυστρία και Τσεχία για παράδειγμα. Πολύ, μπορεί να γίνει και μια θαυμάσια συνεργασία για τις προτεραιότητες. Και το άθο 6, και το άρθρο 6 να αναφερθεί επίσης βιώσιμες μεταφορές και βεβαίως να περιληφθεί ρητά και ο τουρισμός. Αυτά για την ώρα. Και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ. Έχουμε την κυρία Πέτρα εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή του γνωμοδότηση και φυσικά χαιρόμαστε για την υποστήριξή σας σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία και για τα επιμέρους στοιχεία της, αλλά και για την δημιουργία ενός ενιαίου για την, για την ε, επέκτασή της σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Σε ό,τι αφορά τις υποδομές θα διευκρινίσουμε το γεγονός ότι και οι επενδύσεις στις υποδομές εντάσσονται το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και θα το προσδιορίσουμε αυτό στον κανονισμό γιατί υπάρχουν κάποιοι ε, χαμένοι κρίκοι στην διασυνοριακή διασύνδεση και αυτό θα πρέπει να το διορθώσουμε. Θα ήθελα να πω δύο λόγια και για τον τουρισμό. Είναι κάτι που πολύ συχνά επανέρχεται στη συζήτηση γιατί ο τουρισμός είναι σημαντικός κλάδος της οικονομίας και νομίζω ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στους ε, στόχους ε, της στρατηγικής του 2020. Οικονομική ανάπτυξη που θα είναι ευφυής, δεν θα περιθωριοποιεί κανέναν και θα είναι και βιώσιμη. Συμφωνούμε πλήρως λοιπόν. Φυσικά χρειαζόμαστε στρατηγική ε, ενημέρωση και αξιολόγηση της χρήσης των κονδυλίων. Γι' αυτό και υπάρχουν κάποιες διατάξεις του κανονισμού που προβλέπουν την στρατηγική έκθεση, την συνοπτική, συνοπτικές εκθέσεις προόδου για τον τρόπο δαπάνης των κονδυλίων από τα κράτη-μέλη για το 2017-2019 και στην έκθεση προόδου που θα υποβληθεί στην Ειρηνή Σύνοδο Κορυφής θα αναφερθούν κάποια στοιχεία αυτής της έκθεσης να σταθώ σε κάτι που ακούσαμε στη συζήτηση, στην ανάγκη του, της συγκέντρωσης των πόρων, της ε, ε, αποφυγή του, κατακερ... του κατακαιρματισμού των κονδυλίων και της διάσπασης ε, σε πολλές δράσεις και εμείς είμαστε υπέρ της συγκέντρωσης, γι' αυτό και έχουμε διατάξεις για θεματική συγκέντρωση, να περιοριστούμε σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, ε, να εστιαστούμε σε λίγες και καλές προτεραιότητες. Σημαντικό τμήμα της έκθεσης. Σας ευχαριστώ κύριε Κόλιτσεκ. έχετε να προσθέσετε κάτι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να προσθέσουμε τίποτα άλλο σε αυτό το στάδιο, γιατί οι συνάδελφοι αντέδρασαν μάλλον θετικά στην πρότασή μου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τις εργασίες προς την ίδια κατεύθυνση και ευελπιστώ ότι και με τη βοήθεια της ε, Χριστίνας, της βοηθού μου, θα προετοιμάσω μια καλή γνωμοδότηση. Νομίζω ότι και το χρονοδιάγραμμα είναι καλό και η προθεσμία για τις τροπολογίες μας επιτρέπει μια έγκαιρη αντίδραση. Ε, δεν ξέρω, ελπίζω να σας ικανοποιεί το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία ε, για τις τροπολογίες 26 Απριλίου. Οπότε θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Μεταφορών στις 30 Μαΐου και στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης τον Ιούλιο έχει προγραμματιστεί η ψηφοφορία. Επαναλαμβάνω, η διορία για τις τροπολογίες στην Επιτροπή μας ε, είναι 26 Απριλίου. Αυτά να κρατήσετε. Ολοκληρώσαμε την πρωινή μας συνεδρία, αγαπητοί συνάδελφοι, και σε λίγο θα ξεκινήσει και κλεισμένο των θυρών συνεδρίαση των συντονιστών. Σας ευχαριστώ και σας περιμένω με ανυπομονησία στην απογευματινή συνεδρίαση που θα ξεκινήσει με τη συζήτηση της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη. Πρόκειται για κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταφορών και της Επιτροπής Βιομηχανίας που θα ξεκινήσει στις 3. Ένα μικρό διάλειμμα, πεντάλεπτο, για να ξεμουδιάσουμε και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η συνεδρίαση των συντονιστών.